So good morning everybody. A bit exceptionally we have a meeting of the subcommittee on human rights the whole day. Καλημέρα σας. Σήμερα συνεδριάζουμε πρωί και απόγευμα υπό Επιτροπή μας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πέμπτη, δεν ξέρω αν θα έχουμε αρκετό κόσμο. Αρκετά θέματα όμως έχουμε στην ημερήσια διάταξη και θα πρότεινα να κάνω τις ανακοινώσεις Προέδρου λίγο αργότερα όταν ελπίζω θα έχουν έρθει περισσότερα μέλη. και έρχομαι στην ενδιαφέρουσα όσο και επίκαιρη ακρόαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βυρμανία, Μιανμάρ. Αλλά προηγουμένω, ε, σε εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη, θυμίζω ότι θα συζητήσουμε την έκθεση κυρία Αντρικέιν, την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, παρουσίαση για την πρωτοβουλία ΡΕΚΟΜ στα Βαλκάνια, για την Επιτροπή Αναζήτηση και Αποκάλυψη Αλήθεια για τα κλίματα πολέμου και το απόγευμα θα έχουμε ακρόαση σχετικά με την καταπολέμηση τη ατιμορρησία, στο παράδειγμα τη Αργεντινή και πολλέ επισκέψει και σύντομε ανακοινώσει καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα για προβλήματα επίκαιρα και οξέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έρχομαι λοιπόν σημείο 4, ακρόαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βυρμανία Μιανμάρ, εν ώψη των κοινοβουλευτικών εκλογών στις 7 Νοεμβρίου του 2010. Τακτικά μας απασχολεί η κατάσταση στη Βυρμανία. Πρέπει να σας πω ότι απευθύθηκα στην ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο Λέδη Άστον πρόσφατα εν ώψη και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ε, ΟΗΕ και αναφέρθηκα και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Βυρμανία που καλεί ε, στο σεβασμό και υποστήριξη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για μια διεθνή ερευνητική επιτροπή έτσι ώστε να διαπιστωθούν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βυρμανία και στη Βόρεια Κορέα. Είναι μια διαρκής προσπάθεια εξέλιξη αυτή. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους τρεις ε, εκλεκτούς μας ε, προσκεκλημένους ε, στην ακρόαση και θα τους παρακαλέσω να μιλήσουν τρία λεπτά, συγγνώμη, δέκα λεπτά και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς είναι ο κύριος Μπεν Ρότζερς, που εκπροσωπεί μια ε, χριστιανική οργάνωση East Asia Christian Solidarity Worldwide που δραστηριοποιείται στη Βυρμανία και είναι και ο συγγραφέας ενός βιβλίου που πρόσφατα ε, δημοσιεύθηκε για τον ηγέτη ε, του καθεστώτος. Ο τίτλος είναι «Ξεσκεπάζοντας τον τύρανο της Βυρμανίας» και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τι θα μας πείτε. Ε, δεύτερη ε, προσκεκλήμα είναι η κυρία Ζώια Φαν, διεθνής ε, συντονίστρια της εκστρατείας από το Ηνωμένο Βασίλειο της οργάνωσης Berman Campaign UK που παραστέκεται στο λαό της Βερμανίας που υφίσταται τόσο στιγμή καταστολή έχει ξανάρθει στην Επιτροπή μας πέρυσι η τρίτη ειδική ε, προσκεκλημένη είναι η κυρία Ντέμπι Στόταρτ, συντονίστρια του εναλλακτικού δικτύου ΑΣΑΝ για τη Βερμανία και από τη Διεθνή ε, Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναπληρώτρια γραμματέας. Ε, ναι, sorry, next week in Την άλλη εβδομάδα στις Βρυξέλλες θα λάβει χώρα μια σύνδεση κορυφής ΕΣΑΝ αν δεν απατώμε στις 4 και 5 Οκτωβρίου προσπαθώ να προσκαλήσω τις πολιτικές ομάδες να ζητήσουν ε, δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου στη μήνυ σύνοδο του Κοινοβουλίου μας που θα είναι αμέσω μετά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ε, επίκαιρο αυτό και καλή ευκαιρία να ακούσουμε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια θα είναι τα συμπεράσματα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ΑΣΕΑΝ. Ελπίζω οι πολιτικές ομάδες να συνεργαστούν και να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ε, επίσης τη σοβαρή κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα όπως είναι η Βυρμανία, Μιανμάρ. Ε, και τέλος θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρέας Λίστ από τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών ε, Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ε, τον παρακαλέσω να απαντήσει εξ ονόματο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα όμως έχουμε τη μεγάλη τιμή να παρευρίσκεται ο κύριο Ρότζη, τον οποίο και δίνω αμέσω το λόγο. Is this... you can hear me now? <laughs> Thank you very Σας ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση της ε, ακρόασης αυτής σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τη Βερμανία και για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας απευθύνω σήμερα το λόγο. Η κατάσταση στη Βερμανία από πλευρά ε, πολιτική, ανθρωπιστική και κοινωνική και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν ε, δύσκολη τα τελευταία χρόνια, τρία χρόνια, αλλά από το 2007 την ειρηνική ε, διαδήλωση των βουδιστών μοναχών που κατεστάλλει η βία έχει επιδεινωθεί πολύ. Είχα την ευκαιρία να ε, μεταβώ στα σύνορα Ταϊλάνδης ε, Βυρμανίας και να δω πολλούς πρόσφυγες Καρέν που έφυγαν νύχτα από τη χώρα και με πήγαν και σε οριζόνες τη νύχτα γιατί είναι πολύ δύσκολο να επισκεφτώ ένα καταβλισμό. Εκεί συνήντησα έναν άντρα, Καρέν, που η ιστορία του είναι συμβολική για τη σημερινή Βερμανία. Είναι συνομήλικός μου, 35 ετών και έχει χάσει και τα δύο του πόδια από ναρκή όταν έψαχνε στη ζούγκλα για τροφή. Ε, στην καλύβα του από μπαμπού, μέσα στο σκοτάδι, τον... Ε, ε, ε, κυνήγησαν οι ε, Ταϊλανδοί και ε, ο στρατός της Βυρμανίας και μου είπε ότι χρειάστηκε να φεύγω όλη μου τη ζωή, φεύγω για να γλιτώσω από το στρατό της Βυρμανίας. Είναι η Βυρμανία ένα καθεστώς πάρα πολύ στιγνό, ένας από τους χειρότερους δικτάτορες κυβερνάει, ο στρατηγός Θαν Σουέ είναι σε κατάταξη τρίτος μετά τον Κιμ Γιονγκ Ιλ και τον Μουγκάμπε ως παγκόσμιος τύρανος. Έχει δείξει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει καμία συμπόνια για το λαό του και ε, ε, ο μόνος του σκοπός είναι να διατηρηθεί στην εξουσία ε, εκείνος και να διατηρήσει τα πλούτη της οικογένειάς του. Η Βυρμανία από τότε που ανέλαβε με πραξικόπημα ο είναι, έχει ε, κυβερνηθεί από σειρά ε, στρατιωτικών καθεστώτων. Ο Ταν και ο ίδιος στρατιωτικός ήταν ε, αφού στην αρχή της καριέρας του ταχυδρομικός. Μην νομίζετε όμως ότι δεν είναι έξυπνος άνθρωπος, εφής σε πολλέ περιπτώσει έχει εμφανιστεί πάρα πολύ πονηρό, γιατί με χειραγώγηση έφτασε στην εξουσία και τη διατήρησε. Η στρατιωτική του εκπαίδευση είναι στο ψυχολογικό πόλεμο και η τακτική του διέρηκε βασίλευε και το έχει χρησιμοποιήσει ε, σε μεγάλο βαθμό και μεγάλη αποτελεσματικότητα ε, και ε, με τους αντιπάλους του εντός χώρας και προς τη διεθνή κοινότητα. Υπό το καθεστώς αυτό η Βερμανία έχει καταταγεί από τις πιο φτωχές, πιο διεφθαρμένες και πιο ε, κατασταλτικές χώρες και καθεστώτες στον κόσμο. Εκτός ε, ε, από ε, τις ιδιότητες που έχουν όλοι οι δικτάτορες ο Τάγκσο είναι και πάρα πολύ εθνικιστής και αδιάλακτος απέναντι σε οποιαδήποτε εθνοτική μειονότητα που δεν είναι Βυρμανή. Αυτό ξεκίνησε από την Ανατολική Βυρμανία μεταξύ των Καρέν, Καρένι και Σαν και ο βιασμός χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα και συστηματικά ως όπλο πολέμου και η καταναγκαστική εργασία είναι ρουτίνα κακοποιούνται, βασανίζονται ή σκοτώνονται οι χωρικοί. Οι γυναίκε, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι έχουν πολλέ φορέ εκτελεστεί εν Είδα μια γυναίκα, γνώρισα μια γυναίκα τη οποία ο, ο άνδρα τη αποκεφαλίστηκε, ενώ μια άλλη τη οποία είχαν βγάλει τα μάτια του παιδιού τη και είχαν κόψει τα χείλη του και τη μύτη του. Χρησιμοποιούνται σαν αρκαλιευτέ οι χωρικοί. Από το 1996 πάνω από 3.500 χωριά έχουν καταστραφεί στην Ανατολική Βυρμανία, μια κλίμακα καταστροφή που μόνο τον Ταρφούρ έχει αντίστοιχη. Πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπων έχουν εκτοπιστεί και έχουν ξεφύγει στη ζούγκλα ή σε στρατόπεδα επανα... επανεγκατάστασης. Όταν επιτίθεται ε, ο στρατό στα χωριά, πολλέ φορέ αφήνει νάρκες γύρω-γύρω για να μην μπορούν να επανέλθουν οι χωρικοί στα χωριά του. Γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο που σας είπα, ο οποίος είχε χάσει τα πόδια του και σας δείχνει αυτό πόσο μεγάλα είναι τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει κατά της ανθρωπότητας στη Βερμανία και ο ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής, της, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει καταλήξει το ίδιο συμπέρασμα. Στη Δυτική και Βόρεια Βερμανία, το καθεστώς του Τάνσουε εξακολουθεί τις βιαιότητες κατά του τοπικού πληθυσμού. Γνώρισα μια γυναίκα από τη φίλη Κατσίν κοντά στην στα σύνορα της ε, Κίνας που είχε, βία, που είχε βιαστεί και είχε, ε, είχε, απαγχω, είχε ε, στραγγαλιστεί από στρατιώτες. Προσπαθήσαν να τη σκοτώσουν αλλά επεβίωσε. Άλλοι έχουν αντιμετωπιστεί με αντίστοιχους τρόπους. Και παρά το γεγονός ενώ το καθεστώς του Ταν Σουέν εξακολουθεί να καταπιέζει τους βουδιστές, ε, το κάνει το ίδιο και με φυλές όπως η Σαν, Μον και Ρακάν. Δείχνει λοιπόν και μία προκατάληψη κατά των χριστιανών και των μουσουλμάνων, των μη βουδιστών και χειραγωγή και θρησκεία για πολιτικούς λόγους. Οι χριστιανοί Τσιν αναγκάστηκαν να κατεβάσουν τους σταυρούς που είχαν βάλει σε βουνοκορφές σαν σύμβολο της ε, πίστη τους και να εξαναγκάστηκαν σε καταναγκαστική εργασία για το σκοπό του κράτους. Οι Ροχίνγκα που είναι μουσουλμάνοι είναι ένας από τους πιο καταπιεσμένους λαούς στην Βυρμανία. Αν θυμάμαι καλά, χθες το Αμερικανικό Κογκρέσο πέρασε το πρώτο ψήφισμα σε σχέση με την κατάσταση των Ροχίνγκα στην ε, Βιρμανία. Δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα παρά το γεγονός ότι έχουν ζήσει για γενιές στη Βυρμανία. Αντιμετωπίζουν μεγάλες ε, δυσκολίες για πρόσβαση στην ε, παιδεία και μετακίνηση μέσα στη χώρα υπήρξαν στο, είδα στον Μπαγκλαντές ε, λιποτάκτες από το βερμανικό στρατό που μου το επιβεβαίωσαν. Μου είπαν ότι βρισκόμαστε στην, στο χείλο της εξαφάνισης της Αλάος. Ήθελα να πω μερικά πράγματα ακόμα για το Ταν Σουέ. Και είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζει αυτό η διεθνή κοινότητα και να προσπαθήσει να καταλάβει ποιο είναι αυτό με τον οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχει μια πατριαρχική αντιμετώπιση και αυτό φαίνεται και από τη στάση του εναντίον της Aung η οποία είναι σε κατοίκον κράτη τα τελευταία 25 χρόνια. Ο Τάουσι έχει αρνηθεί να προχωρήσει σε διάλογο μαζί της και τις λίγες φορές που έχουν συναντηθεί η στάση του είναι ότι σαν νεότερη από αυτόν και γυναίκα δεν έχει το δικαίωμα να τον επικρίνει. Ένας ε, παρατηρητής ο οποίος ήταν παρόν είπε ότι κατά την άποψή του ο ρόλος της Αγσούξη είναι απλώς να φτιάνει τσάι και να κάνει ευχάριστη να κάνει ευχαριστά συνομιλητικά σχόλια. Ο Ταν Σουί βλέπει τον εαυτό του σαν μια σύγχρονη ε, εκδοχή του πολέμαρχου στην αρχαία Βυρμανία. Και αυτό οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας ε, πρωτεύουσα τη Νάπιντο που στα βερμανικά σημαίνει η πόλη των βασιλέων γιατί υπήρχε αυτή η παράδοση να φτιάνει ο κάθε βασιλιάς καινούργια πρωτεύουσα. Επομένως δεν πρόκειται για ένα άτομο το οποίο θεληματικά θα παραδώσει σε κάποιον άλλον την εξουσία, ούτε κάποιο ο οποίο μπορεί να ακούσει τη λογική. Η μόνη γλώσσα που ξέρει, σαν στρατιωτικό, είναι η γλώσσα τη βία. Ο εμπειρογνώμη για τη Βιρμανία Μπέρτιλ Λίντνερ, λέει ότι είναι τελείω μάταιο να περιμένει κανεί ότι οποιαδήποτε μορφή διαπραγματεύσεων με αυτή την κυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει σε έστω και ελάχιστε αλλαγέ και δημοκρατικοποίηση. Είναι ένα τύρανο και οι τύρανοι δεν διαπραγματεύονται την αποχώρησή του. Τούτου λεχθέντος, παρά την άποψη άλλων αναλυτών, όταν Ταν Σουέ και οι άλλοι στρατηγοί στη Βερμανία μπορούν να αντιδράσουν στην πίεση της διεθνούς κοινότητας. Αλλά η πίεση αυτή μέχρι στιγμής δεν ήταν σωστά στοχευμένη και ήταν σχετικά χλιαρή. Μια σωστή στρατηγική η οποία θα συνδυάζει ε, στεναρά μέτρα κατά των στρατηγών και παρουσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Βερμανία είναι απαραίτητη. Με τον τρόπο αυτό, οικονομικά και διπλωματικά μέτρα, με, αν έχουν τη σωστή στόχευση και εφαρμογή, μπορούν να έχουν ένα σωστό αποτέλεσμα στη Βερμανία. Κλείνω με μερικές σκέψεις για το τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την απόψή μου. Πρώτον, θα πρέπει <clears throat> να απορρίψει τις στιμένες εκλογές του Νοεμβρίου που δεν έχουν καμία νομιμότητα και πρέπει να κάνει σαφέ προ το καθεστώ τη Γερμανία και προ τη διεθνή κοινότητα ότι αυτέ οι εκλογέ είναι απλώ ένα τρόπο διαιώνιση του στρατιωτικού καθεστώτο επί τη βάση ενό νέου συντάγματο το οποίο δεν έχει καμία νομιμότητα και δεν είναι τρόπο αλλαγή. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να απαλύνει τι κυρώσει στη Βερμανία μέχρι ότου υπάρξει ουσιαστική αλλαγή. Τα τωρινά μέτρα θα πρέπει να διατηρηθούν μέχρι ότου υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα όπως η απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και το τέλος των επιθέσεων κατά των αμάχων πολιτών καθώς και η δημιουργία ενός διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης των δημοκρατικών κινήσεων και των εθνοτικών ομάδων. Δεν πρέπει να υπάρξει λοιπόν αμοιβή του καθεστώτος αυτού για τα εγκλήματά του. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εργαστεί ενεργά ώστε να πιέσει τον ΟΗΕ να ξεκινήσει μια συζήτηση υψηλού επίπεδου για τον τριμερή διάλογο που ανέφερα προηγουμένω προ την Εθνική Συμφιλίωση. Τέλο, η τελική μου σύσταση και αυτή που νομίζω ότι θα είναι πιο άμεση σε επίπεδο δράση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τι ε, εκκλήσει για να σταματήσουν τα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα που έχει κάνει το καθεστώ του Τάνσουε πάνω από 12 χώρες έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για τη σύσταση του ΟΗΕ να ξεκινήσει μια επιτροπή έρευνας για την έρευνα ακριβώς αυτών των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Αυτό περιλαμβάνει πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη όθηση προ αυτή την κατεύθυνση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο ζήτησε να υπάρξει μια τέτοια ερευνητική επιτροπή. Είναι καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να προσθέσει τη φωνή της στη φωνή αυτών που θέλουν τέλος στην ατιμορρησία στην Βυρμανία. Μόνο έτσι ο Ταν Σουέ θα μπορεί να πιεστεί να σταματήσει αυτά που έχει κάνει στο λαό της Βυρμανίας τόσα πολλά χρόνια. Ελπίζω ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παίξουν ενεργό ρόλο να παροτρύνουν τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ύπατη εκπρόσωπο για να υποστηρίξει αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Ρότζερς και για τις ε, τέσσερις συστάσεις που κάνατε στο τέλος. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ενεργό και υπεύθυνο ρόλο σε τα πλαίσια αυτής της ε, Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής. Ίσως ε, θα μπορούσε να μας πει και κάποια πράγματα το Συμβούλιο, αν υπάρχει κάποια κίνηση από πλευράς του προς αυτήν την κατεύθυνση. Η επόμενη είναι η κυρία Ζώγια Φάν η οποία θα κάνει και αυτή μια παρέμβαση από την Perma ε, Campaign UK. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που οργανώνετε αυτή την ακρόαση και που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας μιλήσω σήμερα. Κυρία Πρόεδρε, τρία χρόνια πέρασαν από την εποχή που κατέφυγαν στους δρόμους οι βουδιστές μοναχοί ζητώντας αλλαγή, ζητώντας το τέλος στρατιωτικής δικτατορίας, ζητώντας δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Οι βουδιστές μοναχοί αντιμετώπισαν τις σφαίρες και τα όπλα. Πολλοί συνελήφθησαν, πολλοί βασανίστηκαν και πολλοί παραμένουν ακόμα στις φυλακές σήμερα. Ορισμένοι δεν κρύβονται. Για να αποφύγουν τη διεθνή πίεση, τα μέλη του καθεστώτος ε, ετοιμάζουν αυτές τις ε, ψεύτικες, τις ε, στιμένες εκλογές. Αυτές οι εκλογές θα επιβάλλουν ένα σύνταγμα που θα νομιμοποιήσει το στρατιωτικό καθεστώς χωρίς δημοκρατία, χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς δημοκρατία και ελευθερία για τους ανθρώπους της Βρυμανίας και δεν θα επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν του δημοκρατικού κινήματος ε, Αούν Σαν παραμένει σε κατοίκον περιορισμό. Εδώ και 15 χρόνια είναι σε τέτοιο περιορισμό. Αυτό είναι κατά παράδοση βεβαίως του ε, διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, περίπου 2.200 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βυρμανία βασανίζονται. Δεν, υπάρχουν καθόλου, δεν υπάρχει καθόλου ιατρική περίθαλψη για αυτούς αποστέλλονται σε φυλακές σε μακρινές περιοχές και κανένας δεν μπορεί να τους επισκεφθεί. ούτε καν από την οικογένειά τους. Το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης έχει απαγορευτεί, η λογοκρισία, η καταστολή υπάρχει και έχει αυξηθεί και η δικτατορία επίσης ε, απειλή ότι θα σταματήσει την κατάπαυση του πυρός με τις διάφορες εθνοτικές ομάδες, κάτι που θα οδηγήσει σε ανθρωπιστική κρίση ε, στη Γερμανία. Με βάση το Σύνταγμα, ο πρόεδρος θα πρέπει να έχει στρατιωτικό, να είναι στρατιωτικός. Και επίσης ο υπουργό, ε, βασικά η Υπουργεία θα πρέπει να είναι στα χέρια των στρατιωτικών, όπως παραδείγματος χάρη το άμυνας, το εσωτερικό κτλ. Αυτό το Σύνταγμα, με αυτές τις εκλογές, δεν θα ενδυναμώσει απλώς το στρατιωτικό καθεστώς, αλλά θα εξαλείψει και, την, ε, και τις διάφορες εθνικές ομάδες ε, στη Βυρμανία. Ποια είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν διχασμένες για το θέμα της Βερμανίας και ότι πρέπει να γίνει. Ορισμένες χώρες λένε ότι αυτές ε, οι εκλογές είναι εντελώς στημένες, ότι θα πρέπει να τις ε, καταδικάσουμε, ότι δεν θα επιφέρουν καμία αλλαγή. Αλλά όμως υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που λένε ότι αυτές οι εκλογές θα φέρουν κάποια αλλαγή και ότι θα πρέπει να χαλαρώσουν οι κυρώσεις και θα πρέπει να γίνει μια νέα αρχή. Κυρίες και κύριοι, σας λέω ευθέω ότι δεν θα υπάρξει πραγματική αλλαγή. Δεν υπάρχει πραγματική αλλαγή στη Γερμανία. Το κείμενο εναντίον των εθνικών μειονοτήτων ε, έχουν συνταχθεί και η δικτατορία στη Βερμανία διαπράττει ανθρώπινα, ανθρώπινες παραβιάσεις, ε, ε, σταυρώσεις, βιασμούς, με πολλές μορφές βασανιστήριων, ξυλοδαρμό, εκτελέσεις, αποκεφαλισμό και καταναγκαστικά έργα. Κυρία Πρόεδρε, πάνω από 3.500 θρησκευτικοί ηγέτες έχουν φύγει από τα σπίτια τους τα τελευταία 15 χρόνια. Ακόμη και εγώ έφυγα από την πατρίδα μου λόγω της καταπίεσης. Ε, το καθεστώς ε, τα έχει βάλει με τους αμάχους. Κυρία Πρόεδρε, στην αρχή του χρόνου ήμουνα στη Βυρμανία, συναντήθηκα με μια γυναίκα 24 ετών, ήταν όταν αναγκάστηκε να μεταφέρει βαριά φορτία για τους στρατιώτες του Βυρμανικού στρατού. Το βράδυ τη βίαζαν ομαδικά. Την υποχρέωναν να μεταφέρει τις προμήθειές τους, τα εφόδια τους και όταν ο πατέρας προσπάθησε να την ε, υπερασπιστεί για να σταματήσει αυτός ο ομαδικός βιασμός, ε, επιτέθηκαν στον πατέρα τους και όλοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Επίσης συναντήθηκα με μια οικογένεια η οποία ε, είχε ξεφύγει από τους όλμους του στρατιωτικού καθεστώτος και από, τους, από τις βόμβες του. Ένα παιδί από αυτήν την οικογένεια, μαζί με τους φίλους του, πήγε σχολείο στο σχολείο ακριβώς αυτό, ε, το σχολείο αυτό βομβαρδίστηκε, το παιδί τραυματίστηκε και δύο ε, μέρες μετά πέθανε. Οι στρατιώτες γνωρίζουν που κρύβονται οι άμαχοι, οι απλοί πολίτες. Ήξεραν που βρίσκονταν αυτό το σχολείο. Γι' αυτό ακριβώς πυροβόλησαν. Και μάλιστα εξεράγησαν και όλοι σε αυτό το χωριό. Ένα άλλο άτομο αναγκάστηκε επίσης να μεταφέρει εφόδια του στρατού. Αυτό γίνεται συστηματικά. Το καθεστώς χρησιμοποιεί τον κόσμο σαν σκλάβους. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κάνουν αυτή τη δουλειά. Η Μουμπλό είναι ένας από, μία από αυτούς. Την ανάγκασαν να μεταφέρει μαζί με τα παιδιά της ε, μέσα στη ζούγκλα πολύ βαριά φορτία και να περπατάει τεράστιες αποστάσεις χωρίς να αναπαύεται και χωρίς να τρέφεται σωστά. Τελικά αναγκάστηκε να τραπετεύσει. Τα κατάφερε να τραπετεύσει. Ένα άλλο έγκλημα που διαπράττει το καθεστώς στη Βυρμανία είναι η χρήση των παιδιών ε, στρατιωτών. Όταν ήμουν στα σύνορα με την ε, Ταϊλάνδη, ε, συναντήθηκα με κάποια τέτοια παιδιά που είχαν φύγει, που είχαν τραπετεύσει. Μου είπε ένα παιδί ότι ήταν σε επίσκεψη στους παππούδες του όταν το άρπαξε ο στρατός και του είπε ή θα πας φυλακή ή θα καταταγεί στο στρατό. Ήταν παιδί, δεν ήθελε να πάει στο στρατό αλλά αναγκάστηκε και τον έστειλαν σε διάφορες ε, περιοχές εθνικών μειονοτήτων, ε, αναγκάστηκε να διαπράξει εγκλήματα, προσπάθησε να τραπετεύσει, την πρώτη φορά δεν τα κατάφερε, τελικά τα κατάφερε αργότερα. Μόνο και μόνο επειδή έφυγε από το στρατό θα μπορούσε να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκιση 40 ε, ετών. Καταλαβαίνουμε κυρίες και κύριοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει ό,τι μπορεί με τα πολύ στεναρά ψηφίσματα που έχει περάσει και στο παρελθόν. Υπάρχει και αυτό το ψήφισμα που ζητάει από τον ΟΗΕ να δημιουργήσει μια εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει τα εγκλήματα της δικτατορίας της Βερμανίας. Παρά τα ψηφίσματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρά το ότι ο ειδικό απεσταλμένος του ΟΗΕ ζητάει αυτή την διερεύνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, δεν έχει αποφασίσει ακόμα να υποστηρίξει αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Οι εκλογές που προγραμματίστηκαν για τις 7 Νοεμβρίου, το ξέρουμε σήμερα, δεν θα επιφέρουν πραγματική αλλαγή για τον λαό της Βρυμανίας. Δεν θα επιφέρουν τις αλλαγές που θέλουν και ελπίζουν οι άνθρωποι οι πολίτε της Βυρμανίας. Έχει και ώρα λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπόλοιπη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνε της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα ε, ελπίζουμε να υποστηρίξει αυτή την εκταστική επιτροπή του ΟΗΕ ε, που θα διερευνήσει τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εναντίον του βυρμανέζικου λαού ήγηκε η ώρα η διεθνή κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβουν την πραγματική φύση της δικτατορία στη Βερμανία. Αυτή η δικτατορία αποτελείται, τα στελέχη της είναι στατιωτική. Δεν είναι πολιτική, δεν είναι διπλωμάτες. Δεν θα ανταποκριθούν σε χαλαρά ή ήπια μέτρα, όπως αυτά του ΟΗΕ. Σαράντα επισκέψεις οι απεσταλμένοι του ΟΗΕ έχουν κάνει τα τελευταία 40, ε, τα τελευταία χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπήρξε καμία δημοκρατική αλλαγή στη Βυρμανία. Πρέπει να υπάρξει πιο ισχυρή πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να καθοριστούν και όρια και χρονοδιαγράμματα γιατί χωρίς πραγματική αλλαγή θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για το καθεστώς. Ζητάμε τη διεθνή κοινότητα να αυξηθεί αυτή η πίεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να χαλαρώσει τις κυρώσεις χωρίς να υπάρξουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στη Βυρμανία. Θα πρέπει να υπάρξει στοχευμένη οικονομική πίεση, πολιτική πίεση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη διεθνή κοινότητα. Κυρίε και κύριοι, Ξέρουμε το καθεστώς ούτως ή άλλως θα διοργανώσει τις εκλογέ. Μετά από αυτέ τι εκλογέ όμω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει ένα διάλογο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στη Βιρμανία. Ο ΟΗΕ κατ' επανάληψη ζήτησε να γίνει τριμερής διάλογος. κατορία από τη μία το δημοκρατικό κίνημα υπό την αιγύδα της Αούν ε, Σουκή και των δημοκρατικών εκπροσώπων στην ε, Βυρμανία. Επίσης, ο ΙΕ θα έπρεπε να συναντηθεί με εθνικούς εκπροσώπους ε, των διαφορών μειονοτήτων στην Βυρμανία. Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη πίεση από τη διεθνή κοινότητα, ούτως ώστε να το δημοκρατικό κίνημα, οι εκπρόσωποι των διαφόρων μειονοτήτων και η δικτατορία να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να κάνουν πραγματικέ διαπραγματεύσει για να επιλυθεί το πρόβλημα τη Βερμανία. Ο λαό τη Βερμανία ζει μέσα σε φοβερή φτώχεια. Έχουν ανάγκε οι οποίε δεν καλύπτονται. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Βερμανία καθώς και μεγαλύτερη διασυνοριακή βοήθεια. Υπάρχουν περίπου 500.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν μέσα στη Βερμανία, γιατί μπλοκάρεται η κίνησή τους από τη δικτατορία. Μόνο μέσω των συνόρων, των εξωτερικών συνόρων της Βερμανίας μπορούν να μετακινηθούν. Μέσω της ε, ε, Ταϊλάνδης, της ε, Ινδίας και άλλων γειτονικών χωρών. Και της Κίνας βέβαια. Αυτό το που θέλει το δημοκρατικό κίνημα στη Βερμανία είναι μια πραγματική δημοκρατία. Όχι μια ψεύτικη δημοκρατία. Μέσω ενός τριμερούς διαλόγου Κάτι που επιζητεί και επιδιώκει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλε χώρε. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να διπλασιάσει τι προσπάθειέ τη για να πείσει και να υποστηρίξει τον ΟΗΕ να, για να προωθήσει την ιδέα αυτή του τριμερούς διαλόγου. Για να υπάρξει επίσης εθνική συμφιλίωση η οποία τελικά θα οδηγήσει σε δημοκρατία. Θέλουμε μία ομοσπονδιακή Βιρμανία με όλες τις φυλές μας, με όλες τις θρησκείες μας, ε, όλοι θα πρέπει να είναι ίσοι, άντρες και γυναίκες. Από όλες τις φυλές θα συνεχίσουμε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την, α, της διεθνούς κοινότητας προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούτε λοιπόν ότι όλοι οι παρόντες εκτιμούν και υποστηρίζουν την ισχυρή έκκληση που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια θέση στεναρή και να τη διατρανώνει. Σας ευχαριστώ και για τις υπόλοιπες προτάσεις για τη διασυνοριακή βοήθεια και για την υποστήριξη του τριμερούς διαλόγου. Βεβαίως, στο τέλος θα κάλεσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει και να απαντήσει στις προτάσεις και στα αιτήματα, ιδιαίτερα ότι αφορά τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα όμως να δώσω το λόγο στην κυρία Ντέμπι Στόταρτ από το εναλλακτικό δίκτυο ΣΕΑΝ για τη Βυρμανία να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Κυρία Στόταρτ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Θα ήθελα εισαγωγικά, κυρίες και κύριοι, να πω ότι είμαι από τη Μαλαισία και ζω στην Ταϊλάνδη και εργάζομαι για τη Βερμανία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι κάθε φορά που κάνουμε πρόοδο στα πολιτικά δικαιώματα, στα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΑΣΕΑΝ. Υποστηρίζουμε ε, και τις χώρες ε, ΑΣΕΑΝ. Οι χώρες ΑΣΕΑΝ έχουν χαλαρώσει, γιατί έχει χαλαρώσει η Ευρώπη. Αν σκληρύνει τη στάση της Ευρώπη, θα είναι και πιο σκληρή η στάση των ασιατικών χωρών. Δηλαδή, ουσιαστικά η νοοτροπία στην περιοχή μας και η στάση των κυβερνήσεων εξαρτάται κατά 65% από την Ευρώπη, γιατί προσανατολίζονται στην αντίδραση της Ευρώπης. Αν εσείς κάνετε λιγότερα, θα κάνουν και εκείνοι λιγότερα. Εγώ λοιπόν εδώ θα ήθελα σήμερα να τονίσω τα σοβαρά προβλήματα στη Βυρμανία, τα οποία επιδεινώνονται. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να ε, δώσει την πρόφαση στην Ασία για να μην ε, δράσει στη Βυρμανία. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το Σύνταγμα και τον εκλογικό νόμο και τις εκλογές. Σύμφωνα με αναλύσει μας, η διεξαγωγή των εκλογών, ο εκλογικός νόμος και τα βασικά στοιχεία στο Σύνταγμα είναι οι ρίζες ε, της σύγκρουσης της πολιτικής και της οικονομικής κρίσης στη Βυρμανία ε, κατόπιν παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όλα αυτά έχουν οξυνθεί και επιδεινωθεί από τον Νοέμβριο του 2007. Είναι σκανδαλώδη, εξωφρενική εκλογική νόμη που ορίζουν ότι τα κόμματα θα πρέπει να αποβάλουν, να διαγράφουν τους ηγέτες τους όταν κρατούνται στη φυλακή αν θέλουν να συμμετέχουν στις εκλογές. Επίσης, ε, καταδικάζονται ε, πρόσωπα μέχρι και σε κάθε 20 ετών ε, με την πρόφαση ότι παρακολύουν τις εκλογές. Και απαγορεύονται οι ε, πολιτικές συγκεντρώσεις ε, ε, ανθρώπους που θέλουν απλώς να φέρουν τη σημαία τους, της χώρας τους. Επίσης, πάνω από 2.000 πολιτικοί κρατούμενοι έχουν αποκλειστεί από τις εκλογές. Και πολλοί εξ αυτών ήταν πολύ ε, αξιόλογοι και θα ήταν εξαιρετική πολιτική αν τους είχαν επιτρέψει να συμμετέχει. 93 χρόνια φυλάκιση έχει καταδικαστεί ένας ηγέτης των ΣΑΝ. Ένας νέος επίσης ε, καταδικάστηκε σε 104 χρόνια πέρυσι τον Ιανουάριο γιατί μοίραζε φυλάδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το καθεστώς αυτό έχει αφοσιωθεί στο να βεβαιωθεί ότι η πολιτική αυτοί κρατούμενοι ε, να μην έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν όχι σήμερα σε εκλογές, ούτε σε επόμενες ζωές με τόσα χρόνια που έχουν καταδικαστεί. Αν ε, κοιτάξουμε λοιπόν εδώ τα στοιχεία που έχουμε, θα διαπιστώσουμε ότι το 90 η έδρες ήταν 492 και το 2010 έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των εδρών, ωστόσο είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό εκείνο των κομμάτων και των προσώπων που επιτρέπεται να συμμετέχουν στις εκλογές για όλες αυτές τις θέσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν διαπιστώσουμε ότι το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν και να επιλέγουν την κυβέρνησή τους είναι πραγματικά θεμελιώδες δικαίωμα. Και από τα στοιχεία αυτά διαφαίνεται ότι στη Βυρμανία δεν συμβαίνει αυτό. Το δικαίωμα του λαού να ασκεί τα δημοκρατικά του δικαιώματα, να αποφασίζει ποιο θα τον εκπροσωπεί, παραβιάζεται και περιορίζεται σημαντικά. The of the Δεν θα μπω ε, στις διατάξεις του συντάγματος που ευνοούν τη σύγκρουση. Απλώς θέλω να σας πω ότι ε, εδώ σας δείχνω ένα χάρτη για το ε, που ενδέχεται μέσα στον επόμενο χρόνο να ξεσπάσει ε, πόλεμος. Είναι το πορτοκαλί περιοχές που οι κοινότητες καταπιέζονται, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και θέλουν να προστατεύονται. If we Λοιπόν, αν θέλουμε να μειωθούν οι συγκρούσει και να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να ε, παρατηρήσουμε τον επόμενο χάρτη, ο οποίο δείχνει ότι 3.000 χωριά στερήθηκαν την ευκαιρία να κάνουν εκλογές. Η Εφορευτική Επιτροπή δύο εβδομάδες και λιγότερο τώρα δήλωσε ότι συγκεκριμένα 3.014 χωριά δεν θα κάνουν εκλογές. Και βλέπετε πώς αντιστοιχεί ο χάρτης αυτός που σας δείχνω. Ε, αντιστοιχεί στις έφλεκτες περιοχές. Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα η Φορευτική Επιτροπή αρνήθηκε απέρριψε τις υποψηφιότητες 14 εκπροσώπων εθνοτήτων. Είναι πάρα πολύ ε, μεγάλη οι περιορισμοί ε, των εκπροσώπων διαφόρων εθνοτήτων ε, και υφίστανται καταπιέσεις και εγκλήματα. Φέτος από το Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο έχουμε αποδεδειγμένα διαπιστώσει ότι είχαμε 15 θανάτους, ε, εκτελέσεις χωρίς ε, δίκες, ε, με, ε, εκτοπισμούς, εξορίες. Τουλάχιστον 14 ε, κρατούνται αυθαίρετα, 8 περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής βίας και συστηματικές διώξεις της, των μειονοτήτων Ρεχίνγκα που είναι μουσουλμάνοι εδώ κρατώ και μόλις έλαβα μία έκθεση που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες, τη Δευτέρα συγκεκριμένα. Και η έκθεση αυτή αφορά την καταναγκαστική στρατολόγηση παιδιών τους τελευταίους μήνες στη Νότια Βερμανία. Σε ε, μικρά χωριά από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο έχουν στρατολογηθεί τουλάχιστον 40 παιδιά με τη βία για στρατιωτικούς σκοπούς από το στρατό της χώρας, SPDC. Σε ένα και μόνο χωριό ανάγκασαν 40 ε, μάχους να ε, καταταγούν σε ένα παραστρατιωτικό τμήμα που ελέγχεται από το στρατό και από τους 40 τα 15 ήταν παιδιά. Τους τελευταίους 6 μήνες σε άλλα μέρη της χώρας Τουλάχιστον δύο παιδιά στρατολογήθηκαν ε, με τη βία ως παιδιά στρατιώτες και ένα άλλο παιδί που αρνήθηκε, δολοφονήθηκε ε, από τους στρατιωτικούς. Λοιπόν, για το λόγο αυτό έχω έρθει ενώπιόν για να σας πω και να επαναλάβω ότι τώρα περισσότερο από ποτέ είναι επίκαιρο και σημαντικό η Ευρώπη να δείξει στεναρή στάση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Εάν η Ευρώπη δεν το πράξει αυτό και ανταυτού ε, τηρήσει στάση αναμονής, βλέποντας και κάνοντας, ε, κινδυνεύουμε να δούμε τα χειρότερα σενάρια, που είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και το φρικτό ενδεχόμενο η εντός εισαγωγικών εκλεγμένη βουλή στη Βυρμανία που κυριαρχεί ο στρατός να ε, εγκρίνει ε, τον πόλεμο και τις ε, βίες και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα που κατοικούν άλλε εθνότητες. Βέβαια, αν δεν γίνει πόλεμος, μπορεί και πάλι να μην αλλάξει η κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι μια χούφτα άνθρωποι στο κοινοβούλιο έχουν το θάρρος της γνώμη τους και τα λένε αυτά, δεν έχουν την εξουσία να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί δεν υπάρχει αρκετή εξωτερική πίεση. Ακόμα και αν θέλουμε να υποστηρίξουμε εκείνους που ε, αντιστέκονται στη Χούντα, θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε από την Ευρώπη με στεναρή στάση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Βερμανία. Θα ήθελα να σας πω και άλλα πολλά, αλλά οι δύο προλαλήσαντες νομίζω είπαν ε, όσα έπρεπε να υποθούν. Ε, προσυπογράφω και συμφωνώ απολύτως με όλες τις στάσεις. Αυτό χρειάζεται τώρα η Βυρμανία και επίσης θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα θύματα των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου έχουν το δικαίωμα στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη και στη γνώση ότι είναι στο πλευρό τους η διεθνής κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και προσιλωμένη πλήρως στο σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων. Και κάτι άλλο ακόμα πιο σημαντικό να τα λέμε αυτά δημόσια, να τα εννοούμε σοβαρά για να το καταλάβει και το καθεστώς. Τέρμα πια τα εγκλήματα. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ και εγώ. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Στόταρντ. Ακούσαμε πολύ σαφείς συστάσεις ε, και κλήσεις ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακούσουμε τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θέλουμε να καλωσορίσουμε και δύο ομάδες στη συνεδρίασή μας. Υπάρχει μια ομάδα διερμηνέων από διεθνείς οργανισμούς που κάθονται πίσω-πίσω. Είμαι τιμή μας που είσαστε παρόντες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίασή μας. Ξέρω ότι εκπροσωπείτε σημαντικές οργανώσεις όπως το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Ιουγκοσλαβία, τη Διεθνή Οργάνωση Υγείας και τα λοιπά. Έχουμε επίσης μια ομάδα ακτιβιστών από τη Γερμανία που τους έφερε εδώ το Γραφείο για τη Γερμανία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπος αυ... αυτής της ομάδας θα ήθελε να πάρει το λόγο για ένα-δύο λεπτά. Ναι, βλέπουμε ένα χέρι, έχετε το λόγο για μια σύντομη δήλωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μας προσκαλείτε για να πάρουμε το λόγο σήμερα. Είναι τιμή να βρισκόμαστε εδώ. Φτάσαμε από τη Βερμανία χθες μαζί με τους συναδέλφους μου και προσωπούμε την κοινωνία των πολιτών που δραστηριοποιείται στη Βρυμανία. Ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να πω πολύ σύντομα κάποια βασικά πράγματα. Παρά την προσπάθεια των διεθνών οργανώσεων, παρά την προσπάθεια για την προστασία των πολιτών, ε, δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα. Υπάρχει συνεχής προσπάθεια. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στη συμμετοχή του λαού παράλληλα με την προσπάθεια οικοδόμησης θεσμών που ξεκινάει από πάνω. Αν θέλουμε να υπάρξει μια πραγματική δημοκρατία πρέπει να ενεργοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών. Ε, δημοκρατία σημαίνει ενεργοποίηση των πολιτών. Πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι για να διαμορφώσουν το μέλλον του θα πρέπει και εκείνο να, να Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βοηθήσει την ανάπτυξη της δημοκρατίας και της κοινωνίας των πολιτών στην Μιενμάρ. Γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξει τις οργανώσεις αυτές που δίνουν δύναμη στο λαό. Τα κινήματα της κοινωνίας των πολιτών που στηρίζουν τις αξίες της, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και που κάποια μέρα θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και την ειρήνη στη δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι και, μια ώρα για να στήριξετε περισσότερο τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Βοηθήστε ούτως ώστε να δημιουργηθούν μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, και να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν διάφορα φόρουμ ε, όπου θα συναντώνται διάφορες οργανώσεις κοινωνία των πολιτών, των γυναικών, των νέων. Αυξήστε την ανθρωπιστική βοήθεια και πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ζητήστε ανεξαρτησία για τον τύπο. Ζητήστε περισσότερη κατάρτιση και εκπαίδευση. Και συμμετοχή με ειρηνικά μέσα. Επίσης σας ε, καλούμε να ζητήσετε διάλογο με τις αρχές, να συνεχίσετε να ασκείτε πίεση, να βοηθήσετε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Να υπάρξει θεσμική μεταρρύθμιση, να υπάρξει μεταρρύθμιση του τομέα της ε, άμυνας, Νομίζω ότι η προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω και, και από κάτω προς τα πάνω θα πρέπει να γίνουν παράλληλα, ούτως ώστε να υπάρξει πραγματική δημοκρατία στη Βυρμανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στις Βρυξέλλες και Ξέρω ότι πολλοί από εσά θα συμμετέχετε στο Φόρουμ ε, Συνεργασία Ευρώπη-Ασία στα πλαίσια του ΑΣΕΑΝ. Και το θέμα τη Βυρμανία ενδεχομένω να συζητηθεί και σε αυτό το πλαίσιο. Νομίζω ότι έχει φτάσει τώρα η ώρα να στραφούμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών ε, ε, Σχέσεων. Παρακαλώ. Τώρα με την νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας ελπίζω ότι θα έχουμε πιο ενωμένη θέση. Θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις της ΥΠΑ της εκπροσώπου, της Λέδης Άστον. Ε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις προηγούμενες παρεμβάσεις. Δεν θα σχολιάσω τα επιμέρους σχόλια και παρατηρήσεις ε, για τις φρικαλαιότητες στη Βυρμανία. Αν δείτε την γενική κατάσταση της οικονομίας, την έλλειψη σωστής διατροφής των παιδιών, ε, δύσκολη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, ε, τα πράγματα μιλάνε από μόνο τους νομίζω. Νομίζω ότι είναι και η ώρα η ύπατη εκπρόσωπος να κάνει κάτι, γιατί ούτω ή άλλως ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν θα μακρηγορήσω για την, σε ό,τι αφορά την ανάλυση μας για τις εκλογές. Αρκεί να κοιτάξετε την ανάλυση του, της ομάδας των φίλων του Γενικού Γραμματέα Μπαν Κιμούν που συναντήθηκαν τις τελευταίες μέρες ε, υπάρχουν διάφορες χώρες, η Κίνα, η Ινδία, χώρες ε, ΑΖΕΑΝ, που είπαν ότι θα πρέπει να δούμε με θετικό μάτι την κατάσταση, γιατί υπάρχει μια διαδικασία αλλαγής, αλλά υπάρχει μια αίσθηση απογοήτευσης, δεν μπορεί να μας διαφύγει αυτό. Γνωρίζω ότι ακόμη και εκπρόσωποι της Ιαπωνίας έχουν τεράστιες εκπροσώπ, ε, αμφιβολίες για τις εκλογές. Πώς γίνεται να γίνουν πραγματικές ε, εκλογές αν οι περισσότεροι εκπρόσωποι είναι φυλακισμένοι και η ίδια η Άννου Σανσουκή. Η κατάσταση λοιπόν είναι ζωφερή. Τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι να δούμε αυτές τις εκλογές και άκουσατε διάφορες απόψεις για αυτό το θέμα. Ο ένας τρόπος είναι να θεωρήσουμε ότι ούτως ή άλλως είναι προβληματικές, τιμένες και ότι δεν έχουν νόημα. Αυτή είναι η άποψη πολλών κρατών μελών και το διατρανώνουν και προς τα έξω. Και είναι μία άποψη που είναι προϊόν δύσκολων αποφάσεων και την ίδια άποψη έχει και η Άουν Σαν και το κόμμα της. γι' αυτό αποφάσισε να μην συμμετάσχουν, να μην συμμετάσχουν σε εκλογέ. Υπάρχουν και άλλοι όμω, όπω ξέρετε, που λένε παρά τις δυσκολίες, παρά τις ζωφερές προοπτικέ, αξίζει να κάνει κανεί μια απόπειρα Μήπως υπάρξουν κάποια στοιχεία, κάποιες αλλαγές, κάποια πρόοδος και βγούμε λίγο από αυτήν την πολύ δύσκολη σημερινή κατάσταση. Η Ντέμπι είπε ότι αυτή είναι η άποψη και κάποιων κρατών μελών. Αλλά πιο σημαντικό είναι η ίδια η άποψη πολλών ανθρώπων της Βυρμανίας, όχι μόνο κάποιων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που όπως αναφέρθηκε προωθούν αυτή την ιδέα, αλλά με βάση κάποια τελευταία ε, στοιχεία, περίπου 260 υποψήφοι κατεβαίνουν και είναι εκπρόσωποι των λεγόμενων δημοκρατικών κομμάτων αντίπαλοι της κυβέρνησης. 30 αυτά τα κομματα κατεβασουν κατεβάζουν περίπου 250-260 υποψηφίους. Μέσα σε ένα πλαίσιο, η εκστρατεία τους γίνεται μέσα σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο. Το κόστος της καταχώρησής τους είναι τεράστιο, αλλά υπάρχουν και περιορισμοί για τις ε, συγκεντρώσεις τους, την εκστρατεία τους, την προεκλογική κτλ. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς προεκλογική εκστρατεία σε, μια, σε ένα πλαίσιο που η Χούντα είναι πανταχού παρούσα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να υποστηρίξουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να τους αγνοήσουμε, να αγνοήσουμε τις απόψεις τους. Η γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τις δικές τους προσπάθειες μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο. Θα ήταν δύσκολο να υπάρξει, όταν, αν υπήρχε αντίθεση ανάμεσα σε αυτούς τους ε, ε, αντιπάλους της κυβέρνησης, σε περίπτωση που οι ΜΕΝ λέγανε ότι πρέπει να υπάρξει συμμετοχή και οι άλλοι όχι. Εμείς δεν θα χαλαρώσουμε την ε, υποστήριξή μας. Νομίζω ότι η διαφωνία μεταξύ των αντιπάλων της Χούντας θα ήταν προς όφελος της Χούντας. Θα περιμένουμε μέχρι να λάβουν χώρα ε, οι εκλογές και θα αναλύσουμε μετά τι συνέβη. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος γι' αυτό. Νομίζω ότι στις αρχές του 2011 θα μπορέσουμε να αποφανθούμε για τη σημασία των εκλογών. Όπως είπε η Ντέμπη, το θέμα δεν είναι μόνο πόσο, πόσες έντρες θα πάρουν οι υποψήφοι της αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι ποιος θα έχει τα βασικά υπουργεία ε, και κυρίως ε, τι πολιτικές θα υπάρξουν. Ε, αν θα υπάρξουν διαφορές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τον τρόπο διαχείρισης οικονομίας κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να δοκιμαστούν στην πράξη. Υπάρχει ελπίδα, αν τα δούμε όλα συνολικά, ότι η κυβέρνηση θα χαλαρώσει την πρόσβαση και ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή από τις διάφορες οργανώσεις στην όλη διαδικασία. Πολλοί μίλησαν για την ανάγκη να αλλάξει η ανθρωπιστική κατάσταση, να δοθεί βοήθεια στο λαό της Γερμανίας. Μία αποστολή της ΕΚΟ θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες και ένα από τα πράγματα που θα εξετάσει θα είναι κάτι συνομιλίες με τις αρχές, η δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης στην Ανατολική Βυρμανία προς τα σύνορα με την Ταϊλάνδη, πρόσβαση δηλαδή των μελών της αποστολής αυτών των περιοχών. Ε, είναι περιοχές που δεν έχουμε επισκεφθεί ποτέ στο παρελθόν, δεν μπορέσαμε να έχουμε πρόσβαση. Τώρα, ας πάω στο θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Να σας υπενθυμίσω ότι τον Απρίλιο το Συμβούλιο των Υπουργών συζήτησε το θέμα της Βιρμανίας, η Μιενμάρ, και το Συμβούλιο διατράνωσε την υποστήριξη το, στην Ban ki αλλά ε, επικύρωσε και την έκθεση Κιντάνα. Θέλω να τονίσω ότι παρά την άποψη που ακούσετε ότι είναι ήπια η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Γερμανία, σε κάθε φόρουμ θέτει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, συνομιλώντας με τις γερμανέζικες αρχές. Η, η κυρία Άστον συναντήθηκε στη Μαδρίτη ε, με εκπροσώπους των αρχών, αλλά και με άλλες ε, γειτονικές χώρες, Κίνα, Ινδία και με διάφορες χώρες ΑΖΕΑΝ ε, πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να παραμείνει ψηλά στην ατζέντα και στις ολομέλειε Ολομέλειες ΑΖΕΑΝ, αλλά και σε διμερείς συναντήσεις που ο πρόεδρος Μπαρόζο και ο πρόεδρος Φαν θα έχουν ε, με χώρες και ηγέτες ε, ΑΖΕΑΝ. Παραμένει λοιπόν ψηλά στις προτεραιότητε μας και της Γκλέδης Άστον. Γνωρίζω από την πείρα μου ότι είναι πολύ δύσκολες κάποιες μακρές διαπραγματεύσεις ε, για τέτοια θέματα, διαπραγματεύσεις που είναι ατέρμονες. Εμείς θα κάνουμε πάντως προσπάθεια και κάνουμε προσπάθεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, τι θα γίνει εφ' εξής. Οι εμπειρογνώμονες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν ήταν σε επαφή με ορισμένους από εσά για το θέμα της εξεταστικής αυτής επιτροπής. Για μας η λιδία λήθος είναι τι θα αλλάξει στη χώρα αυτή. Καλές είναι οι δηλώσεις, οι βαρύγδουτες θα είναι δηλώσεις. Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι που θα αλλάξει τα πράγματα στη Γερμανία. Υπάρχουν θέματα χρόνου, χρονοδιαγράμματος δημιουργίας υποστήριξης ύπαρξης υποστήριξη σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες. Η Γερμανία δεν είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, γι' αυτό θα πρέπει το θέμα αυτό να τεθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ε, υπάρχουν και άλλα θέματα, να μην τα αναφέρω όλα. Πάντως δεν έχουμε αποκλείσει αυτό το θέμα. Ε, και ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, με τον Κέρτ Κάμπελ από τις Ηνωμένε Πολιτείες είχαμε επαφές και ο Κέρτ Κάμπελ είπε ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν αποκλείσει τίποτα. Θα κοιτάξουν ε, τι θα γίνει μετά τις εκλογές τον Νοέμβριο και το πώς θα προχωρήσουμε. Επομένως, συζητάμε θέματα χρονοδιαγράμματος, πώς μπορούν να δημιουργηθούν εκλογικές πώς μπορούν συγγνώμη, να δημιουργηθούν συμμαχίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τέτοια θέματα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα προκύψει από αυτές τις εκλογές και αν η νέα κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει κάτι διαφορετικό. Πάντως, να είστε σίγουροι ότι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό εκ του σύνυγκης. Να επανέλθω σε λίγα θέματα. Συμφωνώ με τον Μπεν για την σημασία και την πρωταρχική σημασία ιδίω που έχουν οι προσπάθειες του ΟΗΕ. Οι προσπάθειες διαλόγου του Κέρτ Κάμπελ και μια προσπάθεια διαλόγου σε υψηλό επίπεδο που προσπαθούμε να προωθήσουμε ε, δεν σημαίνει ότι είναι προσπάθειες υποβάθμισης των, ε, του τι γίνεται σε επίπεδο ΙΕ. Εμείς θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά δεν θα πρέπει ο κόσμος μας, οι άνθρωποι που δουλεύουν επί τόπου, να δίνουν ε, λανθασμένα μηνύματα. Πρέπει να έχουμε μια προσεκτική προσέγγιση για τις ακυρώσεις ε, τώρα. Δεν πρόκειται να αρθούν οι κυρώσει. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να άρουμε τι κυρώσει μετά τι εκλογέ. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα αλλάξουμε καν την κοινή θέση. Ούτε καν θα το συζητήσουμε αν δεν υπάρξουν απτά στοιχεία για θετικέ εξελίξει στη Βιενμάρ. Παραμένουν λοιπόν οι κυρώσει Και σε καμία περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει τάση για χαλάρωση των, κυε... κυρώσεων. Συμφωνώ με αυτά που είπε η για την ΑΖΕΑΝ. Ήταν ατυχής αυτή η αναγγελία των ε, Αμερικανών για τον ενισχυμένο διάλογο με τις αρχές της ε, Γερμανίας. Δώσαν ένα μήνυμα ίσως στην αρχή ότι θα γίνουν πιο χαλαροί, πιο ήπιοι απέναντι στο καθεστώς, αλλά το διόρθωσαν μετά. Δύο χώρες ΑΖΙΑΝ, δεν θέλω να ονομάσω, χάρηκαν πάρα πολύ που δηλώσαμε ότι θα χαλαρώσουμε. Μην ξεχνάτε συνάδελφοι ότι πρέπει να πιέσουμε τη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη πολύ έντονα. Γιατί είναι χώρες που έχουν κάποια οικονομικά συμφέροντα με τη Μάρ και μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα. Στι επόμενε συναντήσει, στην Σύνοδο Κορυφής ΑΖΕΑΝ θα στείλουμε σαφή μηνύματα για το τι περιμένουμε από την ΑΖΕΑΝ τις επόμενες εβδομάδες πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Κυρία Χάουτελα, νομίζω ότι μου δώσατε αρκετό χρόνο από τις απόψεις μου, μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο γενικά για το θέμα της Τα Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τινέσπη. Μιλήσατε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι θέλουμε να έχουμε μία ε, ενιαία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως εξακολουθούμε να βλέπουμε ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν μία άποψη και κάποια άλλη μία άλλη. Είναι πάντοτε λίγο δύσκολο για μας να μην μαθαίνουμε τα ονόματα των κρατών μελών που ανήκουν στα διάφορα, στις διάφορες ομάδες. Υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει με αυτή την προσπάθεια δημιουργίας μιας κοινή εξωτερικής πολιτικής. Εγώ θα ήθελα να ξέρω πάντως ποιοι πιστεύουν τα μεν και ποιοι τα δε. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γκόμες και βεβαίως ε, όποιος άλλος θέλει μπορεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, και εγώ ήθελα να πω ότι Είμαι υπέρ ε, του να είναι η Βυρμανία η υψηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάστασή του το 1988. Προσπάθησα να έχουμε την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε μια επιτροπή που είχε δημιουργηθεί για αυτό το λόγο. Από τότε... Προσπαθώ στην Ασία, στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, το 2002 κατάφερα μάλιστα πολλές φορές να πάω στην ε, Βιρμανία... Προσπαθώ όσο μπορώ να προωθώ το ζήτημα αυτό και πραγματικά θαυμάζω τους ανθρώπους που ζουν εκεί γιατί καταφέρνουν να έχουν μια καθημερινότητα παρά το γεγονός ότι η βιαιότητα της δικτατορίας είναι πολύ μεγάλη. Το 2000 συμμετείχα στην πρώτη ε, εις βάθος ενημερωτική συνεδρίαση που οργανώθηκε για το θέμα αυτό, προσπαθήσαμε να οργανώσουμε κάτι πιο περιορισμένο για την Βυρμανία στην Ασία. Και βεβαίως είχαμε ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό ε, και στο Κοινοβούλιο. και περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όταν ε, ο κυκλώνας έπληξε την ε, ε, Βυρμανία και με τόσο εγκληματικό τρόπο το αντιμετώπισε η δικτατορία της Βυρμανίας και η παγκόσμια κοινότητα δεν έκανε τίποτα. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ καλά είναι τα λόγια, αλλά δεν είμαστε καθόλου αποτελεσματικοί στις πράξεις. Βέβαια τα πράγματα στο παρελθόν δεν ήταν καν όπως αναφέρονται τώρα. Δεν υπήρχε ε, τόσο μεγάλη διάσταση απόψεων και τώρα το πρόβλημα είναι η Κίνα. Επαναλαμβάνω, η Κίνα. Ας δει κανεί τι κάνει η Κίνα για να αποφασίσει ποιος ε, συμφωνεί με τι και από ποια μεριά, σε ποια μεριά τάσεται. Δεν είναι μόνο θέμα βερμανία, είναι και θέμα Κίνας. Εγώ ήμουν από αυτού που αγωνίστηκα να συμπεριληφθεί στο τελευταίο ψήφισμα η ανάγκη συνέχισή των συστάσεων ε, του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα εγκλήματα πολέμου. Ήταν επίσης μια σύσταση και του προηγούμενου εισηγητή του ΟΗΕ για το θέμα αυτό. Και πραγματικά είναι φοβερό το ότι δεν έχει συμβεί τίποτε. Και ο ΟΗΕ έχει ευθύνη. Ο ΟΗΕ είναι αυτός που ε, επέτρεψε να κάνει η Κίνα ό,τι θέλει και επέτρεψε και η Ευρωπαϊκή Ένωση το, το επιτρέπει. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ να ζητήσει από τις Ηνωμένε Πολιτείες να συμμετέχουν και εκείνες ε, για να ανταποκριθούμε επιτέλους ε, σε σχέση στις ευθύνες που έχουμε για τα εγκλήματα πολέμου. Πρώτα απ' όλα βέβαια πρέπει και η Κίνα να συμμετέχει. Και η Κίνα ενδιαφέρεται για την εικόνα της στη διεθνή κοινότητα διαφορετικά. Δεν νομίζω ότι θα είχε αφήσει την ε, παραπομπή της ε, περίπτωσης ε, της υπόθεσης του Μπασίρ να περάσει έτσι από το Συμβούλιο Ασφαλείας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό και ευχαριστώ και τους ομιλητές μας. Είναι γεγονός ότι η ΑΖΕΑΝ είναι σημαντική και εγώ πιστεύω ότι η ΑΖΕΑΝ θα είναι πάντοτε η ποιότερη στην προσέγγιση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη ήπια στην προσέγγιση της, η ΑΖΕΑΝ θα είναι ακόμη ποιότερη. Οπότε πρέπει και η ΑΖΕΑΝ να αναλάβει τις της και ειδικότερα η Ινδονησία που είναι ο μεγάλος παίκτη στην Ασία. Είναι πάρα πολύ σημαντική δημοκρατική χώρα η οποία αν συμμετέχει στις διαβουλεύσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, για μια σωστή προσέγγιση, είμαι απολύτως βέβαιη ότι και η Ινδονησία θα μπορούσε να είναι και αυτή πιο δραστήρια στον τομέα και θα μπορούσε να ε, πείσει και τους υπόλοιπους εταίρους της ΑΖΕΑΝ. Επίσης πιστεύω και χαίρομαι που εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανέφερε αυτό ότι δεν θα μειώσουμε τις κυρώσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι οι κυρώσεις μπορεί να μην δουλεύουν πολύ καλά, γιατί δεν είναι ο σωστός τρόπος να αλλάξει η πολιτική κατάσταση. Αυτό πρέπει να γίνει σε επίπεδο ΙΕ. πρέπει να γίνει. και από την πλευρά να ειδωθούν όλα από την ε, οπτική γωνία των ποινικών, των εγκληματικών ε, δράσεων χρειάζεται η ενίσχυση όλων των μέσων των οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όταν πήγα στη Βυρμανία το 2002 είδα ότι η αντιπολίτευση έκανε το εξής λάθος. Νομίζω ότι έκανε πολλά λάθη, ειδικότερα σε σχέση με το οικονομικό πλαίσιο. Όμως έχει αλλάξει η ε, κατάσταση και ίσω θα έπρεπε να δούμε όλες τις διόδους που υπάρχουν για να βοηθήσουμε τη Βιρμανία, ειδικότερα όλους όσους ε, εργάζονται υπέρ τη δικαιοσύνη ε, και τη ισότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ. Thank you. And... Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις παρουσιάσεις Νομίζω ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την κατάσταση και να μην δεσμευτούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί η δραματικότητα της κατάστασης στη Βυρμανία είναι τέτοια που δεν μπορεί παρά να δημιουργείται μια συμπόνια μέσα μας, ακούγοντας όλες αυτές τις μαρτυρίες. Και πρέπει νομίζω να συνειδητοποιούμε πραγματικά το, την ανάγκη για αλλαγή, για δημοκρατία στη Γερμανία. Εκφράζω λοιπόν την αμέριστη αλληλεγγύη μου και σας δηλώνω διατεθειμένος να κάνω ό,τι μπορώ για να συνεισφέρω να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Η συνάδελφος που μίλησε πριν, μίλησε για την ευθύνη της Κίνας. Υπάρχει μια συστηματική δράση η οποία φτάνει στα όρια της αιμονής από πλευράς Κίνας για άμεση πρόσβαση στους φυσικούς πόρους της Βερμανίας. Γι' αυτό η Κίνα λοιπόν βγαίνει από την ε, ευθεία οδό και παίρνει την παρακαμπτήριο για να ορμήξει πάρα αυτά στις, στους φυσικούς πόρους. Δεν κοιτάει κατάματα κανέναν και τελικά στηρίζει κυβερνήσεις ε, που είναι καθαρά δικτατορικές. Φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο να πετύχει συμφωνίες και μάλιστα γρήγορες συμφωνίες ε, προς το συμφέρον της όταν δρά με αυτόν τον τρόπο. Τίθεται λοιπόν εδώ ένα πρόβλημα και μάλιστα θέλω να το θέσω και ως προς κάτι άλλο. Εμείς από πλευράς μας τι δράση θα προωθήσουμε. για να προωθήσουμε ένα άλλο δικαίωμα του ανθρώπου. Βλέπουμε ότι οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Το ξέρουμε. Πρέπει γι' αυτό να διατρανώσουμε ένα θεμελιώδες δικαίωμα. την πρόσβαση στους φυσικούς πόρους των ανθρώπων που ζουν στη Βυρμανία και των μελλοντικών γενεών. Νομίζω ότι μια δράση προς αυτήν την κατεύθυνση για αυτό το δικαίωμα στους φυσικούς πόρους μπορεί να διαφυλάξει και ζωντανή την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει πραγματική, βιώσιμη, δημοκρατική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόντι. Δεν ζητάει κανένας άλλος βουλευτής το λόγο. Εδώ και τα μέλη της ε, Νοτιοανατολικής Ασίας ε, είναι συνήθις πρακτική ε, εντάσσουμε και γεωγραφικές αντιπροσωπείες στις συνεδριάσεις μας. Ε, νομίζω λοιπόν ότι τρεις, επίσημοι, τρεις ειδικοί προσκεκλημένοι μας ε, θα μπορούσαν να πάρουν το λόγο για λίγα λεπτά για να αντιδράσουν. Άκουσα κάποιες ιδέες από ευρωβουλευτές που έχουν δουλέψει πολύ για το θέμα της Μιανμάρ ότι Συχνά τα αιτήματά σας δεν είναι συγκλίνουν και δεν είναι πολύ καθαρά. Αν κατάλαβα καλά, ε, υπόθηκε ότι ήταν ατυχές να σταλεί ο ειδικό απεσταλμένος, ο κύριος Φασίνο, ε, στη Βυρμανία. Νομίζω ότι δηλώσατε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσατε λοιπόν να το σχολιάσετε. Θα μπορούσε να ξεκινήσει πρώτος ο κύριος Ρότζερς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ευχαριστήσω ε, τους συναδέλφους για όλα τα σχόλια που έγιναν και ειδικότερα ότι δεν θα υπάρξει μείωση των κυρώσεων όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι να υπάρξουν σοβαρές αλλαγές. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα ζητήματα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη σύσταση για ερευνητική επιτροπή. Μπορεί να μην άκουσα καλά, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Γκαλέσπη είπε ότι πρέπει να το υποστηρίξει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Κίνα. Από ό,τι κατάλαβα, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να ε, περάσουμε από τη Γενική Συνέλευση, ε, μέσω ψηφίσματος στη Γενική Συνέλευση μια τέτοιου είδους σύσταση και δεν ε, υπάρχει περίπτωση έτσι αρνηση της Κίνας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε και θα έπρεπε μάλιστα να συστήσει κάτι τέτοιο στην ε, Γενική Συνέλευση φέτος όλας. Τώρα, σε σχέση με τις εκλογές, ο κύριος Γκαλέσπη είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιμένει να δει τι θα γίνει στις εκλογές. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό μέχρι ενό σημείου, αλλά νομίζω ότι με τις συγκεκριμένε εκλογές στη Βυρμανία δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί το, το Σύνταγμα του 2008 και ο εκλογικό νόμος του τρέχοντο έτου, ε, δείχνει πάρα πολύ καλά τι έγινε. Ε, ο στρατός 25% των... Ε, ε των πήρε, υπάρχει πλήρης ατιμορρησία για τα εγκλήματα και πολλές ε, εθνοτικές ομάδες έχουν ήδη αποκλειστεί από τη συμμετοχή τους στις εκλογές, οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις... Ε, ε, οπότε το να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Ίσως θα έπρεπε από τώρα να τις καταδικάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φαν. Κύριε Πρόεδρε, 20 χρόνια βλέπουμε ότι η ήπια προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει αποτέλεσμα. Και το ίδιο εκμεταλλεύεται και η Βυρμανία. Ο κύριος Φασίνο έχει την εντολή να φέρει τις χώρες ΑΣΕΑΝ ε, πιο κοντά στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βρεθεί ε, ένα κοινό έδαφος για το πώ θα αντιμετωπίσουν τη Βερμανία. Ενώ ε, αντί να το κάνει αυτό ο κύριος Φασίνο έφερε την Ευρώπη κοντά στην ΑΣΕΑΝ και χαλάρωσε τη στάση της απέναντι στη Βερμανία. Ε, χρειάζεται ενωμένη ε, προσέγγιση υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών για τη Βερμανία που είναι, είναι στρατηγική προσέγγιση ψηλού επίπεδου και ε, και να συμμετέχουν ε, και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στο δημοκρατικό κίνημα της Aung San Suu και άλλοι δημοκράτες της χώρας. Ευχαριστώ κυρία Στότερτ. Ευχαριστώ. Να επαναλάβω ότι όντως μετά τις εκλογές πρέπει να αναλύσουμε κάποια πράγματα. Αλλά από αυτά που είπε ο Μπεν Ρότζερς και οι υπόλοιποι ομιλητές και εγώ, Γνωρίζουμε ήδη εκ των προτέρων τι είναι πιθανό να συμβεί και ήδη πρέπει να ανασκουμποθούμε για δράση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να δούμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, η Κίνα αρχίζει να αισθάνεται τα ίδια προβλήματα με τις χώρες ΑΖΕΑΝ. Αυτό που, που έμαθαν οι χώρες ΑΖΕΑΝ ε, είναι ότι είναι ένας δύσκολος ε, εχθρός το καθεστώς. Και η Κίνα λέει ότι δεν της αρέσει η αστάθεια στη χώρα που διαιωνίζεται από τα σοβαρά εγκλήματα του καθεστώτος. Τώρα θα πρέπει να δείξουμε θάρρος και να διατρανώσουμε τις αρχές μας. Γιατί πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ακόμα και η χειρότερη καταιγίδα μπορεί να αλλάξει τροχιά εάν υπάρξει κατάλληλη δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο για να αντιδράσει γιατί ακούστηκαν πολλές παρατηρήσεις για την ήπια προσέγγιση. Είπατε δύο λόγια για το θέμα των κυρώσεων, αλλά ίσως να θέλετε να αντιδράσετε και στα άλλα σχόλια. Κυρία Χάουταλα, ε, κάποια σύντομα σχόλια, αν μου επιτρέπετε, για τη Γενική Συνέλευση. Το είχαμε σκεφτεί, αλλά θα υπάρξουν και άλλα προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα θέματα. και να μας κάνουν να προτιμούμε το δρόμο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πάντως το έχουμε κοιτάξει, το έχουμε σκεφτεί. Ε, η διαδικασία μας δεν έχει τελειώσει. Είμαστε σε επαφή με τους Αμερικανούς και με άλλες χώρες και δεν έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Τώρα, για τις εκλογές αυτές καθεαυτές. Μπορούμε να πούμε, θα μπορούσαμε ήδη να πούμε ότι είναι στημένες οι εκλογές και δεν έχουν νόημα. Αλλά φοβάμαι ότι αν κάνουμε κάτι τέτοιο, κλείνουμε τα μάτια και δεν τίνουμε χείρα βοηθείας προς τις άλλες ομάδες. Ε, είναι δύσκολε όντω οι εκλογέ, τι ελέγχουν εκ του σύνεγγυ οι στρατιωτικοί, αλλά δεν θέλουμε να αποστρέψουμε το βλέμμα από τι άλλε αυτέ ομάδε ε, ανθρώπων. Αν είναι να προκύψουν από τις εκλογές αυτές. Άλλοι άνθρωποι, πιο έξυπνοι, πιο δημοκρατικοί, διαφορετικοί κτλ. Ε, δεν θα προκύψουν τόσο πολύ από τις εκλογές ε, που ελέγχονται από τους στρατιωτικούς. Μπορεί να προκύψουν όμως κατά τύχη. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι προσωπικότητες θα, προκύψουν μετά τις εκλογές. Θέλουμε λοιπόν να το δούμε αυτό. <coughs> Αλλά Νομίζω ότι θα κάνουμε μια ασφαλή κρίση για το τι συμβαίνει στις αρχές του 2011 και νομίζω ότι και οι Αμερικανοί έχουν αντίστοιχη άποψη με τη δική μας. Στην αρχική μου παρέμβαση παρέλειψα να αναφέρω τον κύριο Φασίνο, ο οποίος κάνει μια δουλειά ορόσημο από τη στιγμή που διορίστηκε από τον τότε, είπα, το εκπρόσωπο κύριο Σολάνα για την διατήρηση τακτικών επαφών με τις χώρες ΑΖΕΑΝ, με την Κίνα, την Ινδία και άλλες ασιατικές χώρες της περιοχής. Και σε άλλες ε, συναντήσεις στο παρελθόν είχαμε επαφές με αυτές τις χώρες, αλλά αυτός είχε έναν συστηματικό ρυθμό ε, επαφής με, αυτούς, με αυτές τις χώρες. Δεν δεχόμαστε την κρίση ότι αυτός με τη στάση του συνεισέφερε σε μια υπιότερη στάση και χαλαρότερη στάση. Όταν εμείς ανακοινώσαμε ότι θέλουμε να υπάρξει μια προσπάθεια υψηλού επίπεδου, οι χώρες Αζιάν θεώρησαν ότι είναι χαλαρότερη εκ μέρους μας, η ποιότερη στάση. Αν δείτε όμως τι λένε οι αξιωματούχοι, οι Ταϊλανδοί και οι Συγκαπουριανοί, Όντω υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι γινόμαστε πιο ήπιοι, αλλά θα πρέπει να τους βάλουμε, να τους διαψεύσουμε απλούστατα. Για την Κίνα. Μην φανταστείτε ότι η Κίνα ε, θεωρεί ότι η Βυρμανία της δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Η Κίνα σκέφτεται τα επενδυτικά συμφέροντά της, ε, την υποδομή για φυσικό αέριο κτλ. Και χρειάζεται διασφάλιση ότι ο Βυρμανέζικος στρατός θα ρυθμίσει κάποια προβλήματα. Παρ' όλα αυτά η Κίνα αισθάνεται αρκετά άνετα αυτή τη στιγμή με την Βυρμανία και το καθεστώς. Είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε συμπεράσματα, λέει η Πρόεδρος. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το να πιστέψουμε στη σημασία αυτών των εκλογών είναι λάθος. Για αυτή την Εξεταστική Επιτροπή για τις Φρικαλαιότητες, Τη ζητάμε γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γνωρίζει κάθε δικτάτορα σε αυτόν τον κόσμο ότι θα έρθει μια μέρα που θα λογοδοτήσει και θα πληρώσει. Περιμένουμε διάφορες χώρες να ενταχθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να προσυπογράψουν αυτή την αρχή της λογοδοσίας. Πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παραμείνει στεναρό και να εξακολουθήσει να πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί αυτέ οι φρικαλαιότητε που ακούσαμε, όπω είπε και ο κύριο Πρόντι, είναι αποτρόπε, είναι σοκαριστικέ. Ακούσαμε πάρα πολλέ ιστορίε ότι τόσο φρικαλές και αποτρόπε που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν ε, επί προσώπου γης. Σας ευχαριστώ κύριε Ρότζες, ε, σας ευχαριστώ για το βιβλίο σας. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα θέλουν να διαβάσουν ε, το βιβλίο αυτό που παρουσιάζει το πραγματικό πρόσωπο των δικτατόρων της ε, Μιανμάρ. Να κάνω σύντομα μερικές ανακοινώσεις που δεν έκανα στην αρχή της συνεδρίασης και μετά θα προχωρήσουμε θα μιλήσει η κυρία Ανδρική Ένε που έχει να προσθέσει κάτι πριν πούμε στη συζήτηση της ετήσιας έκθεσης, της έκθεσης της. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ στρατηγική αυτή η ετήσια έκθεση, ένα εργαλείο για να ασκεί πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετά θα συζητήσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια με τον κύριο Κούκαν. Λοιπόν, εχθές η Επιτροπή Εξωτερικών συνήντησε την κυρία Ρόζαλιντ Μάρσδεν που διορίστηκε η ειδική εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σουδάν και είχα το προνόμιο να τη συναντήσω την προηγουμένη της συνεδρίας. Πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από τη γνώση της, την εμπειρία της, την εμπειρογνωμοσύνη της και πραγματικά και πιο σημαντικό είναι ότι με έπεισε για τη δέσμευσή της και την παρουσία και της αποστολής της θα ενισχυθεί η υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν. Επίσης, συναντήθηκα με τον Άλλη Αγκάπ και τον Απτελμόνι Αγκάπ από το Σουδάν που επίσης επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουν διάφορες επαφές. Πρέπει να πω ότι και εκείνοι ε, έχουν πει ότι εμπιστεύονται πολύ και εμπιστεύουν στην κυρία ε, Μάρσδεν. Να σας πω και δύο λόγια για το Τουρκμενιστάν. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάει τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκμενιστάν. Εχθές η Επιτροπή Εξωτερικών συζήτησε σχέδιο έκθεσης της κυρίας Νικολάη και ήταν ευρεία η συμφωνία ότι η υποεπιτροπή μας θα μπορούσε να αφιερώσει κάποιο χρόνο πριν εγκρίνει την έκθεση της Επιτροπή Εξωτερικών για να εξετάσει πάρα πολύ προσεκτικά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν και πώς θα ε, προωθηθούν και θα υποστηριχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πήραμε λοιπόν την άδεια, αν μου επιτρέπετε, να ε, διοργανώσουμε ειδική ακρόαση για αυτό το θέμα και θα προσπαθήσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας να το ε, γράψουμε στην ημερησία της 14 Οκτωβρίου, πάντα με τη συμφωνία της εισηγήτριας. Ε, πολλοί βουλευτές είπαν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο και πιο προσεκτικά αυτή τη συμφωνία γιατί θα αποτελέσει προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογεί την προοπτική προώθηση και υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επόμενες ε, συμφωνίες συνεργασίας με άλλες χώρες όπου είναι πάρα πολύ ζωφερό το ε, παρελθόντος προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να επηρεάσουμε σοβαρά την υπόθεση αυτή τη συμφωνία που το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει στη διαδικασία της σύμφωνη γνώμης. Και ο κύριο Αλμπερτίνη πρέπει να σας πω συμφώνησε και τον ευχαριστώ για να γίνει αυτή η ακρόαση, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών. Στη συνέχεια. Ε, ε, προσκάλεσα να μιλήσω στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Τυφλίδα, στη Γεωργία, πριν από δύο εβδομάδες ε, πέρασα μια ολόκληρη μέρα μαζί τους και έχει ενισχυθεί απόψη μου ότι πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με τις επιτροπές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συζήτησα κυρίως με τον κύριο Ντίκ Μάρτι που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά σε αυτή την Επιτροπή για πάρα πολλά θέματα ε, για τις παραδόσεις CIA, θα θυμάστε την έκθεση Μάρτι, και την ε, έλλειψη ε, νομικών μέτρων για να καταπολεμηθούν οι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βόρειο Κάφκασο. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να το δούμε και στο μέλλον και θα ήθελα να πω ότι ενδεχομένω θα μπορούσαμε κάποια φορά να συνεδριάσουμε από κοινού. Ξεκινή συνεδρίαση με την Επιτροπή αυτή γιατί έχουμε αντίστοιχα θέματα που μας απασχολούν και διαπραγματευόμαστε ως επιτοπλίστων. Επίση, θα ήθελα να σα πω ότι το Συμβούλιο τη Ευρώπη. ζήτησε να υποστηρίξουμε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης για το θέμα των Ρωμά. Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβούλιο της Ευρώπης. Και εξ όσων γνωρίζω η Επίτροπος κυρία Ρέντινγκ βλέπει ευνοϊκά την ιδέα αυτή τη συνεργασίας. Και πάλι θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να ξέρουμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει πολύ πραγματογνωμοσύνη, γνώση και έχουμε κάθε λόγο να ε, συνεργαζόμαστε, να αποκομίζουμε και εμεί εμπειρίες που θα μας είναι χρήσιμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο, κυρία Αντρική για να συνεχίσει τι ανακοινώσει. Thank you. Thank you, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο θέμα του Αλήμ που είναι γιος του Ιγούρου ακτιβιστή Αλτεγκύρ, ο οποίος κρατείται από το 2006 και βασανίζεται. Σύμφωνα με ανεξάρτητες πηγές ε, της Κίνας, ο Αλή Αμπτελήμ ε, έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και δείχνει ε, σημάδια σωματικής και ψυχολογικής βλάβης. δεν ε, υπήρξε ιατρική βοήθεια που ε, ζητήθηκε και φυσικά ε, φοβάται για τη ζωή του. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να αναλάβουμε άμεση δράση να κάνουμε έκκληση στις κινεζικέ αρχές προκειμένου ο κύριος Αλή Αμπτελήμ ε, να μην βασανίζεται, να μην, να μην ε, γίνεται κακομεταχείρισή του ε, στην φυλάκιση και τουλάχιστον να, του, επιτραπεί η επίσκεψη ενός ιατρού, να υπάρχει ατρική βοήθεια. Αυτό, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντρικίνε. Μπορούμε να γράψουμε μία επιστολή στον πρέσβη βεβαίω. Θα ήθελα να πω ε, συνεχίζοντας αυτά που, αυτό που μόλις μας είπε η Αντιπρόεδρος, είδα ε, για την κυρία ε, Ράντιαν Καντήρ, ε, την επικεφαλής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ιγούρων, ένα πάρα πολύ ωραίο έγγραφο για ένα φεστιβάλ κινηματογράφου στην Πίσκε αλλά δυστυχώς η μετάδοση διεκόπη γιατί θεώρησαν θεώρησε η ασφάλεια ότι δεν επιτρεπόταν ε, να, μεταδοθεί, να μεταδοθούν οι ταινίε. Ε, θεωρούσαν ότι ήταν θέμα ασφαλείας. Τέλος πάντων είδα ε, πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα για το θέμα αυτό και νομίζω ότι πρέπει να μπορέσουμε να, πρέπει να εξετάσουμε και πάλι τα ζητήματα αυτά των Ουιγούρων. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Νάλντι. Ναι, σε σχέση... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε για τους Ουγγούρους. Θα ήθελα να πω, όπως γνωρίζετε, ότι το Παγκόσμιο Συνέδριο όρισε έναν μόνιμο αντιπρόσωπο στις Βρυξέλλες για δύο χρόνια. Νομίζω ότι κάποιοι εξημών τον έχουν συναντήσει και θα είναι χρήσιμο να τον προσκαλέσουμε να μας ε, παρουσιάσει σύντομα ε, το θέμα. Σε μία από τις συνεδριάσεις μας θα ήθελα να πω για την εξαιρετική πρωτοβουλία που ε, αναλάβατε για το Τουρκμενιστάν και τη σχετική ακρόαση. Πάντοτε παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε μέσα να εφαρμόσουμε τις πολιτικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και τις συμφωνίες και τις διαδικασίες, να σταματήσουμε τις συμφωνίες ή να τις συνάψουμε. Είναι γεγονός ένα μέσο, ότι έχουμε επιτέλους ένα μέσο στα χέρια μας, το οποίο βέβαια πρέπει να το μεταχειριστούμε με τη δέουσα προσοχή. Βεβαίως, νομίζω ότι η ακρόαση θα μπορούσε να είναι σημαντική για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ε, πολλά θα εξαρτηθούν βέβαια από τους εμπειρογνώμονες που θα προσκληθούν. Ε, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι επαφές του με τον εισηγητή και νομίζω ότι και αντιπροσωπείες των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ασία θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να πούμε και στους ομιλητές και στους εμπειρογνώμονες που θα προσκαλέσουμε και από την ε, Επιτροπή αλλά και από άλλους ανεξάρτητους οργανισμούς να επιμείνουν στην βελτίωση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν. Αν εγκριθεί βέβαια το θέμα από το Κοινοβούλιο, ή να προσπαθήσουμε πάση περιπτώσει να διαπραγματευτούμε έναν χάρτη πορείας με το Τουρκμενιστάν για γενικές μεταρρυθμίσει και στη συνέχεια, πιστεύω ότι είναι και η καλύτερη ε, προσέγγιση, να περάσουμε στην έγκριση. Να παρουσιάσουν δηλαδή στοιχεία προ τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο. Σα ευχαριστώ κύριε Ρινάλντι για την αφοσίωσή σας και ελπίζω να το δούμε και στην ακρόαση που ελπίζουμε να διοργανώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Ακόμα είμαστε στο στάδιο του προγραμματισμού για τους ομιλητές και στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας παρακαλώ κάντε προτάσεις γιατί δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή όμως να ε, αποζημιώνουμε ε, μεγάλα έξοδα ταξιδιωμακρινά και είναι και ad hoc και ακρόαση και είναι προχωρημένο και το έτος. Σημείο 5. Ετήσια έκθεση λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2009 και πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Η συγκήτρια είναι αντιπρόεδρό μα, μας, ε, κυρία Λάιμα Αντρικιένε, ε, που έχει ε, καταρτήσει ένα σχέδιο έκθεση. Πρέπει να σας πω ότι είναι μία από τις ευκαιρίες που έχουμε πραγματικά να επηρεάσουμε ουσιαστικά τη μελλοντική πολιτική της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι ενδιαφέρουσα η περίοδος με τις νέες σεισμικές αλλαγές που έχουν επέλθει. Κυρία Ανδρικέν. Θα μιλήσω λιθουανικά. Ε, αγαπητή συνάδελφοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Do we have problem? Mr. What's the problem? They say there was no Lithuanian request, which is unusual. Oh. Well, I've been told that no Lithuanian... μου λέγουν ότι δεν προβλέπεται διερμηνία στα Λιθουανικά διότι δεν ζητήθηκε. Δεν είναι πολύ καλό αυτό, αλλά τι θα κάνουμε τώρα. Okay, so θα το ελέξουμε θα, με τις υπηρεσίες. Ζητώ συγγνώμη, μάλλον θα υποχρεωθείτε να μιλήσετε αγγλικά. Θέλετε να ε, μιλήσω αγγλικά. Γιατί εκεί λέει 15 καμπίνα, δεν είναι λιθουανικά. Sorry, we have to continue in English. Uh, uh, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, από την περασμένη Παρασκευή έχετε λάβει το σχέδιο έκθεσης. Δυστυχώς τα αγγλικά και στα μέσα της επομένης εβδομάδος θα έχει μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών έχει οριστεί η 7η Οκτωβρίου, δηλαδή την άλλη Παρασκευή αλλά ήδη πριν από τις θερινές διακοπές στο διευρυμένο Προεδρείο ζήτησα και για τους συναδέλφους και για μένα να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τροπολογίες των προτέρων. Αλλά και περισσότερο χρόνο. Εάν γίνεται θα ζητούσα και θα παρακαλούσα τη Γραμματεία και την Πρόεδρο να αλλάξει την προθεσμία. Να αλλάξει και να παρατείνει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Όχι δηλαδή στις 7 Οκτωβρίου, αλλά τη Δευτέρα, μετά τις 7. Στις 11 το μηνός δηλαδή. Μπορούμε να επανέλθουμε στη συνέχεια, λέει η Πρόεδρος. Αυτό πείτε πρώτα όσο έχετε να πείτε. Λοιπόν, Συζητήσαμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο το 2009. Είναι η ενδέκατη ετήσια έκθεση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Συμβούλιο και Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζουν τι γίνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη δημοκρατία. Τα άλλα δύο θεσμικά όργανα δηλαδή γνωρίζουν και τι λέμε εμείς. Μπορούμε άρα για να πούμε ότι έχει σημειωθεί εντυπωσιακή πρόοδος, ότι έχουμε κατορθώσει να δρούμε πιο γρήγορα <laughs> ε, στην περίπτωση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες ή να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, διότι ο κύριος στόχος όλων αυτών των εκθέσεων είναι η διερεύνηση, η ε, αξιολόγηση και σε ε, ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα και η επικοδομητική κριτική σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία αλλά και κυρίως να απευθύνει τουλάχιστον κάποιες συστάσεις. Την 1η Δεκεμβρίου του 2009 ετέθη σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Μετά από μακρά προπαρασκευαστική περίοδο. Ε, ε, Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη μια οντότητα με μοναδική νομική προσωπικότητα. Και υπόσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί μπορεί να προσυπογράψει την ΕΣΔΑ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά αφορά και τη σχέση μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, τα νομοθετήματα μας, την κύρωση και την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ποιο είναι τώρα το χρονικό πλαίσιο. Η ετήσια έκθεση καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2008 μέχρι το τέλη του 2009. what comes to my mind όταν ε, μιλώ για αυτή την περίοδο, αυτό που κυριαρχεί στο μυαλό μου είναι οι δολοφονίε δημοσιογράφων στη Ρωσία και το Μεξικό, Φερρυπίν. Είναι οι διώξει που υφίστανται στην Κούβα, στη Λευκορωσία, στην Κίνα, ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα γυναικεία δικαιώματα στο Αφγανιστάν, στο Ιράν και όπω ακούσαμε σήμερα και στη Βερμανία. Και Κάτι άλλο, ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα και πολύ ορατό και προβεβλημένο είναι το βραφείο Ζαχάροφ. Κάθε χρόνο έχουμε ε, το λεγόμενο κατάλογο υποψηφίων όπου γνωρίζουμε ότι πολύ περισσότεροι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλους εκείνους που θα πρέπει να γίνουν γνωστοί στη διεθνή κοινότητα και έχουν θυσιάσει πολλά για να υποστηρίξουν τα δικαιώματα κάποιων άλλων. Γιατί ένα μόνο βραβείο Ζαχάροφ έχουμε. Για τη ελευθερία του πνεύματος. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρές και παραμένουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει εμείς να τις καταγγέλουμε και να τις αντιμετωπίζουμε. Βέβαια δεν είμαστε τέλειοι και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο εσωτερικό έχουμε προβλήματα. Ξενοφοβία, ε, ομοφιλοφιλοφοβία και πολλά πολλά ακόμα προβλήματα. μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, άλλα για μας και άλλα για εκείνους. Θα πρέπει πρώτα να ε, τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας πριν ε, βγούμε να κάνουμε συστάσεις σε άλλους πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται ε, και να υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Ε, when I was on this... Κατά την εκπόνηση της έκθεσης μου για την κατάσταση των ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, έλαβα υπόψη μου ε, και τις προκλήσεις ε, της ε, παγκοσμιοποίησης. Μεταξύ αυτών θα ήθελα να σας αναφέρω και την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας. Η διεθνή τρομοκρατία και η καταπολέμησή της μας σωθεί να αναζητήσουμε νέες λύσεις. Πώς να εγγυηθούμε δηλαδή τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτός επίσης και την ασφάλεια των πολιτών μας χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζουμε άλλα ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλη πρόκληση. Η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Εκατομμύρια ε, ανθρώπων πλήττονται από την κρίση αυτή και θα πρέπει και πάλι να ζητήσουμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε και αυτή την πρόκληση και να εγγυηθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών που πλήττονται από την κρίση. Η τρίτη πρόκληση που αναφέρω είναι η κλιματική αλλαγή. Αυτό αφορά ε, κοινωνίες διαφόρων κρατών και θίγονται ε, περισσότερο πιο ευάλωτες ομάδες, κυρίως οι αυτόχθονες πληθυσμοί. Επίσης υπάρχουν συγκριτικά νέες μορφές παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι εννοώ. Τη λογοκρισία στο διαδίκτυο. Ο Ιγούρη, για παράδειγμα. Ο Αντρέας Σουρούτσι, τον Ιούλιο του 2009 Θυμάστε τι έγινε το πρώτο που έκανε η Κίνα ήταν να σταματήσει το ίντερνετ, να το μπλοκάρει, να το φράξει. Και οι bloggers που προσπαθούσαν να ενημερώσουν για το τι γίνεται, ε, καταδικάστηκαν σε ισόβια, μεταξύ αυτών και γυναίκες. Και έχουμε και τα ονόματά τους. έχουν καταδικαστεί ε, σε ισόβια για αυτό το λόγο. Καταλαβαίνετε ότι είναι νέα μορφή αυτή παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και με τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές ως προς το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εργαζόμενοι την εκτισευτή αυτή ακολούθησα κάποιες αρχές. Θα δείτε ότι περιέχει 12 κεφάλαια, έτσι, χωριστές ενότητες. Το πρώτο αφορά την ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το επόμενο είναι τα διεθνή φόρα και η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Άλλο κεφάλαιο ξεχωριστό αφορά το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τον δικό μας ρόλο εκεί πάλι, στη συνέχεια κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί ασχολούμαι ξεχωριστά με διάφορα θέματα. Θανατική ποινή, βία κατά των γυναικών, βασανιστήρια, ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εμπορικές συμφωνίες, ενίσχυση δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις κλπ. Όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι του ΕΛΚ. Και για μένα πολύ μεγάλη σημασία έχει η ελευθερία της θρησκείας και της λατρείας. Γι' αυτό έχω αφιερώσει ξεχωριστό κεφάλαιο σε αυτό και προσβλέπω στην υποστήριξή σας. Το σχέδιο έκθεσης βεβαίως ε, ε, είναι ανοιχτό στις δικές σας υποδείξεις, τροπολογίες, προτάσεις και ε, περιμένω να τις ακούσω. Άλλη αρχή. Νομίζω ότι θα πρέπει να κατονομάζονται χώρες και να διαπομπεύονται. Name and shame. Χώρες που παραβιάζουν τόσο κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο παρελθόν, θυμάμαι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε ετήσιες εκθέσεις και ψηφίσματα όπου αφιερώναμε χωριστά κεφάλαια σε περιοχές ε, ή ακόμα και σε χώρες ε, μεμονωμένες Κίνα, Ρωσία κτλ. Στη δική μου έκθεση αποφάσισα, πώς να το πω τώρα, ε, να μην κατονομάζω έτσι ε, τις χώρες και να τις εκθέτω, αλλά να έχουμε μια γεωγραφική ευρύτερη προσέγγιση. Πώς να το εξηγήσω, δηλαδή. Αναφέρω και χώρες, μην νομίζετε ως παραδείγματα για τις πιο σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς να αφιερώνουν ξεχωριστό κεφάλαιο για μια χώρα. Αυτά νομίζω ήθελα να σας πω εισαγωγικά για τη συζήτηση και περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας και να απαντήσω σε επικρίσεις σας, έτσι ό,τι άλλο έχετε να πείτε. Uh, Ευχαριστώ. πολύ. Δεν με εκπλήσει που η προσέγγισή σας ήταν τόσο συστηματική και καλύπτει τόσο πολύ καλά τα κέρια θέματα για την ε, δική μας συμμετοχή στη σύνταξη της μελλοντική έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της στατικής μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όπως πολύ σωστά είπατε, αφήνεται αρκετό χώρο για τα μέλη της Επιτροπής μας και τις πολιτικές ομάδες να υποβάλουν προτάσεις και με ικανοποιεί ιδιαίτερα η δομή που έχετε δώσει στην έκθεση αυτή. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και οι εξής βουλευτές Χάουτ, Πρόντι, Κίλνεσεν και άλλοι θα λάβουν το λόγο. Ο κύριος Χάουτ πρώτος. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν πρέπει να μας ε, καταδυναστεύουμε τα διαδικαστικά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι νομίζω εντυπωσιακό που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα της ε, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας για ένα θέμα το οποίο στην μέση διάταξή μας εδώ και πολύ καιρό. Αυτό είναι αντιδημοκρατικό. Είναι γενναιόδορη η εισηγήτρια και μπορεί θαυμάσια να εκφραστεί στα αγγλικά, αλλά πρέπει πάντα να έχει το δικαίωμά τη μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο να χρησιμοποιεί τη μητρική τη γλώσσα και εγώ θα διαμαρτυρηθώ στεναρά. Δεύτερον, ξέρω ότι θα επανέλθετε και στο τέλο. έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η πιο σημαντική για μένα έκθεση του έτους. Και το γεγονός ότι ε, θα κλείσει η διαδικασία υποβολής τροπολογιών την επόμενη εβδομάδα χωρίς να είναι διαθέσιμο το κείμενο σε όλες τις επίσημες γλώσσες, αυτό είναι εξοργιστικό. Ίσως το θέμα αυτό λοιπόν θα πρέπει να τύχει μεγαλύτερης προσοχής. Και φυσικά εσείς κυρία Πρόεδρε βέβαια έχετε την ε, εξουσία να πάρετε μια απόφαση για αυτό το θέμα. Αλλά εγώ θα απογοητευτώ ιδιαίτερα να, αν δεν υπάρξει επαρκής χρόνος για να συζητήσει πλήρως η Επιτροπή μας για τα θέματα αυτά, ώστε να μπορέσουν να κατατεθούν οι κατάλληλες τροπολογίες του, του λεχθέντος. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, κυρία Αντρικέινα είναι συνάδελφο εδώ και αρκετό καιρό και η έκθεσή τη είναι ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη και αξίζει συγχαρητηρίων από όλου μα. Είναι μια πολύ καλή βάση εργασία. Η Επιτροπή μα εδώ και πολλά χρόνια προσπάθησε να θεσπίσει μια προσέγγιση για τα ζητήματα αυτά κατά τομής, όχι κατά τομει κατά θέματα περισσότερο, ώστε να υπάρχει εποπτεία τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τόσο να δίνεται έμφαση στο τι γίνεται στον έξω κόσμο. Και προ αυτή την κατεύθυνση έχει την, πλήρη υποστήριξή μα η κυρία Αντρίκενα. Για κάποιε χώρε ίσω υπήρχε ο πειρασμό να προχωρήσει λίγο περισσότερο. Δεν θέλω να την επικρίνω. Όλοι μα νομίζω ότι καταθέτοντα τι τροπολογίε μα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη πειθαρχία, να μην προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη χρειά και το χαρακτήρα τη έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να ακολουθήσουμε την προσέγγιση που έχει υποδείξει η κυρία Ανδρίκενα. Δεν είναι μια έκθεση που αντιμετωπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά χώρε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λέμε στο Συμβούλιο, δεν λέμε στην ύπατη εκπρόσωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα κατάλογο χωρών που θα πρέπει να υποστούν πίεση, χάρη, για να καταργήσουν θανατική ποινή. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια τέτοια προσέγγιση στα ανθρώπινα δικαιώματα. <clears throat> Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία λέει η κυρία Αντρικάινε στην έκθεσή τη, δεν πρόκειται να τα διεξέλθω όλα. Θα σταθώ σε μερικά μοναχά σημεία. Το θέμα τη ε, διαφάνεια. Μετά από την Σουηδική Προεδρία υπήρξε μια κάμψη στα θέματα αυτά διαφάνεια. Είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε την εισηγήτρια για το ζήτημα αυτό για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και εδώ υποστηρίζω απόλυτα αυτά που λέει η συγγήτρια στο σημείο αυτό και επίσης παρομοίως για τις ε, προτάσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών Υποστηρίζω αυτά που λέει η εισηγήτρια για τις κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά τα βασανιστήρια και την ε, προστασία των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως θα έπρεπε να προσθέσουμε και κάποια στοιχεία για το πόσο καλά προχωράει η εφαρμογή αυτών των αρχών. Και εγώ από ό,τι γνωρίζω δεν υπήρξε σημαντική εκπαίδευση προσωπικού για την εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών. Διορθώστε με για το ζήτημα αυτό, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τη νέα εξωτερική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρχει απαραίτητη κατάρτιση των ε, ατόμων που θα είναι σε αυτήν την υπηρεσία σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση, χαιρετίζω αυτό που λέει η συγγήτρια για την ε, συμπερίληψη τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε δύο νέε εμπορικέ συμφωνίε και χαιρετίζω και το γεγονό ότι λειτουργούν οι κοινοβουλευτικέ μα προτεραιότητε στα ζητήματα αυτά Νομίζω ότι εδώ λοιπόν μπορούμε να τονίσουμε ότι τα πράγματα πήγαινε καλά, δεν πρέπει να υπογραμμίσουμε μονάχα τα προβλήματα που υπάρχουν. Νομίζω ότι υπήρξε ένα ποιοτικό και όχι μονάχα ποσοτικό άλμα στα πλαίσια των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν συμφωνώ λοιπόν επίσης για αυτά τα σχόλια που έχετε για το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων συν αυτό το οποίο έγινε με τη Σρι Λάνκα συνδέεται με αυτό το πρόβλημα, ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζει το κατάλογο των χωρών που ανήκουν στη λίστα GS είναι απόλυτα αδιαφανής και δεν μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας στο σημείο αυτό. Και επίσης, σε σχέση με τις τρεις περιοχές καινοτομία που τονίζει η κυρία εισηγήτρια, η ελευθερία της δεσκευτικής συνείδησης, η λογοκρισία στο ίντερνετ κτλ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα την θρησκευτική ελευθερία. Αυτό δεν είναι ένα θέμα μονάχα ενό κόμματο ή κάποιου άλλου κόμματο και το δικό μου κόμμα υποστηρίζει την ελευθερία λατρεία για όλε τι θρησκείε. Αυτό είναι κάτι που πάντα κάνουμε και ελπίζω ότι θα το έχει υπόψη και η κυρία Ανδρικάινα. Επίση, αυτό που λέτε για τη λογοκρισία στο ίντερνετ, κάτι το οποίο δεν είχαμε περιλάβει από ό,τι γνωρίζω τα προηγούμενα χρόνια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εποφελέστε να το υπογραμμίσω. Και επίσης είναι απαραίτητο να δούμε πως κάνει η κυρία Αντρικέινα να δει το θέμα των ε, επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα από την χρηματοοικονομική κρίση. Ελπίζω ότι θα αντιμετωπιστεί και στο μέλλον, στο μέλλον πλήρως το θέμα αυτό. Κάποιες πιο γενικές ε, παρατηρήσεις σε σχέση με τη θέση της ομάδας μας για όλα αυτά. Υπάρχει πάντα μια χρονική υστέρηση. Πάντα μιλάμε για μια χρονική περίοδο πριν από τον διορισμό της Λέδης Άστον ως υπάτου εκπροσώπου. Και αναφερόμαστε λοιπόν σε μια χρονική περίοδο που έχει ήδη ξεπεραστεί γιατί η υποεπιτροπή μας ήδη αρχίζει να σκέφτεται τι θα γίνει με το τρέχον χρονικό διάστημα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, είναι η δουλειά μας να το κάνουμε φυσικά. Και επίσης σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο το Συμβούλιο είναι ο πιστοδρομικότερο ακόμα περισσότερο. Πολλές φορές κοιτάζει μονάχα το παρελθόν και δεν έχει μηχανισμούς βαθμονόμησης, δεν προσπαθεί να παίξει ένα προληπτικό ρόλο και ένα πιο δυναμικό ρόλο. Δεν λαμβάνει υπόψη πολλές φορές τις τροπολογίες που διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως λοιπόν οι ύπατοι εκπρόσωπες και το Συμβούλιο θα ακούσουν περισσότερο αυτά που λέει η κυρία ενα και δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλαμβάνουμε και πάλι τις ίδιες παρατηρήσεις. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη σχέση των εσωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό στον κόσμο τον οποίο, του οποίου απολαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως θα πρέπει να αναφερθεί το θέμα της ε, μετανάστευσης. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια παράγραφος για τις ε, επιπτώσεις σε ανθρώπινα δικαιώματα αυτής της πολιτικής και επίσης για τα θέματα της τρομοκρατίας. Ίσως όμως στον τομέα της ε, μετανάστευσης είναι χρήσιμο να τονίσετε περισσότερο το θέμα αυτό, διότι κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας δόθηκαν διάφορες υποσχέσεις, οι οποίες από ό,τι ξέρουμε τώρα πια δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως. Και επίσης ό,τι αφορά τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τις κρίσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα των ε, εγκλημάτων πολέμου και να τονιστεί αυτό το θέμα στην Κροατία όπου συνελήφθη πρόσφατα ένα άτομο το, για το οποίο είχε ασκηθεί δίωξη και για την ε, Σρι Λάνκα θα έπρεπε να πούμε περισσότερο για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προχωρήσει σε μια πλήρη έρευνα ενδεχομένων εγκλημάτων πολέμου σε σχέση με τη σύγκρουση στη Σρι Λάγκα ε, κάπως απογοητεύομαι σε σχέση με το γεγονός ότι δεν έχουμε αρκετή προβληματική για την έκθεση Goldstein σε ό,τι αφορά τα Παλαιστινιακά εδάφη. Είναι ένα θέμα το οποίο για πολλούς είναι αφιλεγόμενο, αλλά υπήρξε και ένα πολύ λογικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι ίσως μαζί της θα μπορούσαμε να βρούμε μια τροπολογία η οποία να αντανακλά το πνεύμα της, του ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρί να πάρουμε μια μεροληπτική θέση. Είμαι σίγουρος ότι η κυρία Αντρίκενε θα το δεχτεί αυτό σε ό,τι αφορά τις κρίσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτό το χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να πούμε κάτι ακόμα για τη δημοκρατική δημοκρατία του Κονγκό, το οποίο συζητήθηκε βέβαια μόνο την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, αλλά η έκρηξη βία στο Ανατολικό Κονγκό περιλαμβάνεται στη χρονική περίοδο που διαλαμβάνει η κυρία Ανδρίκαινα, επομένω θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη ε, έμφαση στην έλλειψη ικανότητα των διεθνών δυνάμεων να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση. Χαίρομαι επίση για αυτά που λέει στην παράγραφο 74 και το Γουαντάναμο η κυρία Ανδρίκηνα, αλλά ίσω θα πρέπει να έχει μια πιο εχμηρή προσέγγιση όταν λέει για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ουσιαστικά από ό,τι ξέρω μόνο έξι κρατούμενοι έχουν ε, επανέλθει σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία το τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το επίπεδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να θεωρεί ικανοποιητικό έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίω αν θέλουμε να πείσουμε τι Ηνωμένε Πολιτείε να συμπεριφερθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Και αυτό θα μπορούσα να το συζητήσω λοιπόν μαζί τη, λέει ο κ. Άουιτ. Και βλέπω τώρα τι σημειώσει μου. Επίση θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με το σε ποιο βαθμό η ετήσια έκθεση του Συμβουλίου αντανακλά το περιεχόμενο των κοινοβουλευτικών μας ε, εκθέσεων. Δεν ξέρω λοιπόν αν υπάρχει ένα τμήμα στην έκθεση του Συμβουλίου σε σχέση με τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι τέτοιο, πέστε μου. Εάν δεν υπάρχει όμως θα πρέπει αυτό να αναφέρετε κάπου στην έκθεσή σας γιατί αυτό ήταν μια καινοτομία την οποία είχαμε υπογραμμίσει τα προηγούμενα χρόνια και ίσως θα πρέπει να το υπενθυμίσουμε στο Συμβούλιο με ευγενικό τρόπο και πιο γενικά αν θέλετε σχόλια. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση για μένα έχει μεγάλη πολιτική σημασία γιατί είναι ένας μηχανισμός που προωθεί την λογοδοσία του Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας. Είναι υπόλογοι όλοι αυτοί σε εμά για αυτά που έχουν κάνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι μονάχα μια έκθεση που περιλαμβάνει τα δικά μας σχόλια. Είναι μια έκθεση που προωθεί αυτή τη διαδικασία και δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα εμείς έχουμε τονίσει την αρχή ότι πρέπει να λογοδοτεί σε εμά το Συμβούλιο και η Εξωτερική Υπηρεσία. Πρέπει να εργαστούμε όλοι για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή την έκθεση πριν φτάσει στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Comprehensive... Uh, σας ευχαριστώ κύριε Χάουιτ για την uh, πλήρη και εξαντλητική παρουσίασή σας. Ο κύριος Πρόντιχ το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με τα στοιχεία που παρουσιάζονται και πιστεύω ότι είναι μια έκθεση πολύ λεπτομερής. Ευχαριστώ την εισηγήτρια γι' αυτό. Θέλω να κάνω μια προσθήκη μόνο, που πιστεύω ότι είναι απαραίτητη. σε αυτή την απεικόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποιο είναι το πλαίσιο. Κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Το όριο αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Έχει... Και μάλιστα να το λάβουμε υπόψη μας ρητά. Αφού υπάρχει αυτό το όριο των φυσικών πόρων, νομίζω ότι υφίσταται ένα θεμελιώδες δικαίωμα από πλευράς ανθρώπων να έχουν ίση, ισότιμη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους οι σημερινέ γενιές αλλά και οι μελλοντικέ γενιέ. Πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι πρέπει να υποθεί ρητά σε μια έκταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί αυτό προϋποθέτει ότι εάν είναι περιορισμένοι οι φυσικοί πόροι, μην ξεχνάμε ότι είμαστε αλληλένδετοι, αλληλεξαρτώμενοι η μένα τους δε, οι διάφορες χώρες. Και επομένως θα πρέπει συνενετικά να διαχειριστούμε αυτούς τους φυσικούς πόρους. Και να υπάρχει αυτή η εγγύηση ότι κάθε άτομο θα έχει ίση πρόσβαση με τα άλλα στους φυσικούς πόρους. Μην ξεχνάμε επίση και την αρχή τη ε, βιωσιμότητα. Ότι οι φυσικοί πόροι δηλαδή θα πρέπει να εξακολουθούν να υπάρχουν και για τι επερχόμενε γενναίε. Επομένω υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα από αυτό που αναφέρει η παράγραφος 84. Και μην ξεχνάμε κάτι το οποίο μας απασχολεί πολύ συχνά. Μια πειθαρχία σε ό,τι αφορά την εκπομπή των ε, αερίων του θερμοκηπίου. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα για αυτές τις εκπομπές. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει αυτή η θέση ότι πρέπει να υπάρχει και εκεί η συμμεταχείριση. Ακριβώς για να εγγυηθούμε αυτή την αρχή της ίσης πρόσβασης στους φυσικούς πόρους, θα πρέπει να μην ξεχνάμε μία δέσμευση που έχουμε απέναντι στην ατμόσφαιρα, απέναντι στο περιβάλλον ούτω ώστε να εξασφαλιστεί αυτό το θεμελιώδη δικαίωμα για όλου του ανθρώπου, ίση πρόσβαση στου φυσικού πόρου. Πρέπει να υπάρχει αυτό το δικαίωμα για όλου του ανθρώπου που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Αν υπάρχει αυτό το βιώσιμο επίπεδο είναι ε, ένα στόνος ισοδυνάμου διοξιδίου του άνθρωπο, ε, άνθρακα μέσα στον χρόνο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της εφαρμογής ενός δικαιώματος, δηλαδή το δικαίωμα που, έχουμε, που έχει ο καθένας μας στο να εκπέμπει αυτά τα αέρια. Αν θέλουμε να βγούμε από το αδιέξοδο της Κοπεχάγης, προηγουμένως από το Πότσναν και από το Μπαλί, ελπίζω να μπορέσουμε να πούμε κάτι πιο ξεκάθαρο, ίσως στο Κανκούν, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Ε, πρέπει να υπάρξει μια τέτοια ρήτρα, όπως σας τη διατύπωσα, μια ρήτρα ισότητας. Προτείνω λοιπόν να βάλουμε αυτό το γενικό δικαίωμα για την ε, ισότιμη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, κάτι που προποθέτει και το καθήκον να χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους φυσικούς πόρους. Μαζί με τα δικαιώματα λοιπόν μπορούμε να εξετάσουμε και τα καθήκοντα. Ευχαριστώ. Κυρία Κίλιν Νίλσον. Σας ευχαριστώ για αυτή την έκθεση, κυρία Αντρικίενε. Είναι πολύ αποτελεσματική η δουλειά σας. Είναι σημαντική η έκθεσή σας. Το διάβασα στα αγγλικά. Ελπίζω να μου δοθεί ο χρόνος να το διαβάσω και στα γαλλικά. Και να συνεργαστώ με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μου. Γι' αυτό δώστε μας σας παρακαλώ μια προθεσμία για να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Ξέρω ότι πολλά πράγματα έχουν υποθεί και συμφωνώ με πολλά από αυτά που υπόθηκαν και γράψατε. Γι' αυτό που μόλις τώρα είπε ο οικολόγος συνάδελφος, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Φυσικά εδώ και πολλά χρόνια υπερασπίζουμε μια τέτοια προσέγγιση. Ε, δεν θα ασχοληθώ με αυτά, θα ασχοληθώ με θέματα που δεν τα έφτιαξαν οι προαλήσαντες λοιπόν. Καταρχάς, ένα συγκεκριμένο σημείο και θα επανέλθω και με τροπολογία σχετική, έτσι. Για την παράγραφο 57, για τις δολοφονίες. Μου δίνεις... Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε και άλλες χώρες. Νομίζω ότι εστιάζουμε σε πολύ συγκεκριμένες χώρες του, παλιού, του πρώην Σοβιετικού μπλοκ. Θα ήθελα να αναφέρουμε, Φερρυπίν, έτσι θα κάνω και γραπτή τροπολογία, ε, τροπολογία τη Ρουάντα Φερρυπίν. Γιατί ο Αντρέ Ρουίζε Ρενκά, ε, αντιπρόεδρος των ε, Πράσινων, δολοφονήθηκε πρόσφατα. Το κεφάλαιο 15 όπου καλείται τα κράτη-μέλη να υπογράψουν την Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε να προσθέσουμε στον κατάλογο την Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Περιφερειακών και Μειονοτικών Γλωσσών. Νομίζω ότι αν μας δίνατε χρόνο θα κάναμε και άλλες προτάσεις. Αλλά δεδομένου του χρόνου θέλω να επανέλθω σε ένα σημείο που με ενόχλησε. Καταρχά δεν το καταλάβαινα. Το ξαναδιάβασα λοιπόν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε, να ξαναδούμε το κεφάλαιο 31. Εκεί μιλάτε για το θέμα της έκθεσης Goldstone. Goldstein μάλλον. Δεν κατάλαβα τι εννοείται εδώ πέρα. Εγώ τι θέλω να πούμε όμως. Η έκθεσή σας καλύπτει την περίοδο Ιουλίου 2008 με τέλος του 2009. Είναι αδιανόητο λοιπόν σε αυτή την έκθεση να μην μιλάμε για αυτό το γεγονός που κράτησε 22 μέρες 20, 22 μέρες βομβαρδισμών στη Γάζα, αλλά επί 22 μέρες και στο τέλος των 22 ημερών 1.450 ε, Παλαιστίνοι, κυρίως ε, απλοί πολίτες ε, σκοτώθηκαν, 410 παιδιά 104 γυναίκες, 13 Ισραηλινοί επίσης ε, σκοτώθηκαν, όμως ήταν κυρίως ε, στρατιώτες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό το γεγονός, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που συνέβη στη Γάζα. Και η έκθεση Goldstone, Goldstone όχι Goldstein, είναι πολύ σημαντική γι' αυτό. Ε, επίσης θέλω να πω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να δώσει συνέχεια σε αυτή την έκθεση Goldstone, να την παρακολουθήσει, γιατί νομίζω ότι είναι της αρμοδιότητός μας. Ήθελα να το πω λοιπόν αυτό. Θα κάνω και μία τροπολογία γραπτή. Το λέω ήδη προφορικά όμως για να το ξέρετε. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο μιλάτε για τα κατεχόμενα παλαισιακά εδάφη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν επίσης 11.000 κρατούμενοι στις Ισραηλινές φυλακές, εκ των οποίων είναι πάρα πολύ ανήλικοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν το ζήτημα αυτό, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφορούν επίσης και τις δημοκρατίες. Μας λένε, μας λένε συχνά ότι στην περιοχή αυτή υπάρχει μία δημοκρατία. Επομένως, ε, αφού είναι δημοκρατία, μπορούμε να πετύχουμε πολύ γρήγορα ε, κάποια πράγματα, κάποια πρόοδο για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθουμε στο σημείο αυτό για την περιοχή. Ε, η ομάδα μας έχει να σας κάνει και άλλες μικρές προτάσεις και άλλες τροπολογίες. Αν μας δώσετε λίγο χρόνο θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Άλλοι δύο μιλητές θα πάρουν τον λόγο και μετά η εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω κυρία εισηγήτρια γιατί πιστεύω ότι είναι πραγματικά πλήρης και καλή η έκθεσή σας και γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσει κανείς με τέτοια έκθεση όλα τα βασικά θέματα, γιατί ο τομέας είναι πολύ εκτεταμένος. Χαίρομαι που το συζητάμε λοιπόν το θέμα και καλό είναι να εντοπίσουμε τα σημεία που πρέπει να τονίσουμε περισσότερο και κάποια που πρέπει να τονίσουμε λιγότερο. Συμφωνώ καταρχήν με την δομή του κειμένου σας και με τη λύση που βρήκατε για το πώς αντιμετωπίσετε και θα παρουσιάσετε διάφορα θέματα. Θέλω να τονίσω ότι η παράγραφη 2, 3, 4, 5 περιγράφουν τα πιο σημαντικά πράγματα για τον τομέα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι έχουμε τώρα μια νέα θεσμική δομή, ότι έχουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και χάρη σε αυτή την νέα υπηρεσία έχουμε και την ευθύνη βέβαια να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Και εμεί ω Κοινοβούλιο πρέπει να το ζητάμε αυτό. Πρέπει να το ζητάμε στεναρά. Ότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι η βάση αυτή τη υπηρεσία και η κυρία Άστον έχει κάνει αυτή την υπόσχεση ότι θα είναι. Ο πρώτος ομιλητής είπε ότι είναι σημαντικό οι νέοι υπάλληλοι αυτής της υπηρεσίας όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτή την υπηρεσία εξωτερική δράση να καταρτιστούν καταλήλως, ούτω ώστε να σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τονίζεται και περιγράφεται σαφώς ότι υπάρχει μια νέα κατάσταση με την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι έχουμε τη χάρτα, και επίση το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου είναι πολύ σημαντικό για μα. Η κατάσταση αλλάζει για μα τώρα. Ε, η σχέση μα αλλάζει και αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Επίση πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να υπογράψουν και να επικυρώσουν την σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη αλλά και με, την, ε, με τους φορείς που προβλέπει η συνθήκη του ΟΗΕ. Γιατί όλα αυτά απορρέουν από το γεγονός ότι είμαστε συμβαλόμενο μέρος της χάρτας τώρα. Επίσης, ο Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ έχει ανοίξει γραφείο στις Βρυξέλλες, έχει ξεκινήσει τη δουλειά και η εκπροσώπηση αυτή είναι πολύ σημαντική και μας βοηθάει. Χαίρομαι που μιλάτε, που απαριθμείτε τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα, τα πιο σημαντικά δικαιώματα Πρέπει να καταδικάσουμε καταφανώς και να πάρουμε βήματα από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της χρήσης των παιδιών ως ε, στρατιώτες και ως ε, σεξουαλικά εργαλεία. Κάναμε αυτή τη συζήτηση με αφορμή το Κονγκό. Θα κάνω μια τροπολογία επίσης για τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων. Γιατί είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες όπου και αν βρίσκονται, όπου υπάρχει σύγκρουση μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά και οι εθνικές μειονότητες είναι στο στόχαστρο σε περίπτωση που υπάρχει πόλεμος. Αυτά η δουλειά σας ήταν θαυμάσια και σας συγχαίρω. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρέ μου, θέλω να συμφωνήσω με τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Λυπάμαι που ε, δεν μπόρεσατε, κυρία Ανδρική, να μιλήσετε στην ε, μητρική σας. Εδώ στο Κοινοβούλιο υποτίθεται ότι προωθούμε την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία. Λέμε ότι η χρήση της μητρικής γλώσσας είναι σημαντικό θέμα. Η δυνατότητα να μιλάει κανείς στη μητρική του, να εκφραστεί στη μητρική του, είναι κάτι το εκ των όνου κάνευ, το ουσιαστικό. Επομένως, θα πρέπει να εφαρμόζεται και για τους ευρωβουλευτές, όπως και για τους υπόλοιπους πολίτες της Ένωσης. Ας μην μιλάμε τώρα για την ανάγκη μετάφρασης. Είναι σκανδαλώδες το γεγονός ότι δεν έχουμε ε, έτοιμη τη μετάφραση στις γλώσσες μας για να δουλεύουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Αν προσθέσουμε τώρα και την προθεσμία που έχουμε για τις τροπολογίες, νομίζω ότι φτάνουμε στα όρια του απαράδεκτου. αλλά εντάξει, συχνά δουλεύουμε σε σκληρές συνθήκες. Η έκθεση, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντική. Είναι η πρώτη φορά που στα πλαίσια της νέα θεσμική λειτουργίας ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, στο νέο θεσμικό πλαίσιο ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και επομένω θα πρέπει να έχουμε το χρόνο να δουλέψουμε σωστά. Γενικά συμφωνώ με την προσέγγιση της εισηγήτριας. Πολύ σύντομα θα πω κάποια στοιχεία. Ίσως αναφερθώ με, μια διαφορετική απόχρωση. Χαίρομαι για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Επί δεκαετίες ε, ασχολήθηκα με αυτά και πολέμησα για αυτά. Είναι σημαντικό κάπου να μιλήσουμε για αυτά οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Αλλιώς τι νόημα έχει να λέμε ότι υπερασπίζουμε την ε, καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμφωνούμε επίσης ότι θα πρέπει να βάλουμε τάξη στον οίκο μας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε και μια καθολική εικόνα για τα ανθρώπινα και άποψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για το πώς παρουσιάζουμε όμως τώρα τα διάφορα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω να πω κάποια καινούργια πράγματα. Αυτά που στην άλλη δεν θα τα αναφέρω ξανά. Θέλω να παριθμίσω απλώς χίδιν και σύντομα κάποια πράγματα, ούτω ώστε να βάλουμε μια τάξη. Είναι κρίμα που δεν μιλάμε για την πολιτική γειτονία. Την περασμένη εβδομάδα το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Η πολιτική γειτονία είναι οι ε, προτιμησιακέ εταιρικέ ε, συμφωνίε που έχουμε με όμορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτέ τι χώρε θα πρέπει να ειδωθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα για να μην δημιουργήσω προβλήματα. Αυτό που συμβαίνει στη Λιβύη αυτή τη στιγμή δεν είναι αποδεκτό. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τις χώρες του Μαγκρέμπ, για τις χώρες του Μασρέκ και όχι μόνο για αυτές ε, για τις οποίες έχουμε γενικά επικρίσεις και καταγγελίες. Όλες. Θα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την πολιτική του Ισραήλ, για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, την πολιτική της Τινησίας για τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διάφορα παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, τόσο ώστε να έχουμε μια έκθεση πιο ισορροπημένη σε αυτό το τομέα. Ε, Επίση, καταλαβαίνω ότι είναι επικίνδυνο να δίνουμε παραδείγματα. Γιατί όταν δίνουμε παραδείγματα, κάπου δίνουμε έμφαση και άρα δημιουργούμε κάποιε ανισορροπίε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, λοιπόν. Ε, με ποιον τρόπο αναφέρουμε αυτά τα παραδείγματα. Π.χ. Μιλάτε για την ε, κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν. Είναι σκανδαλώδης όντως. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν άπειρες άλλες χώρες όπου η κατάσταση των γυναικών είναι εξίσου σκανδαλώδης με το Αφγανιστάν. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε στο πώς παρουσιάζουμε λοιπόν αυτά τα παραδείγματα. Στη διατύπωση αν θέλετε των παραδειγμάτων. Στη φρασιολογία που χρησιμοποιούμε. Ε, Επίση, είμαι άθεη. Ε, με τη γαλλική έννοια του όρου. Αυτό, παρόλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να προασπίσουμε τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία του να πιστεύει να μην πιστεύει κανείς. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ όλους όσους πιστεύουν σε κάποια θρησκεία και που πέφτουν θύματα εξαιτίας της πίσης τους. Υπό τον όρο θα υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία πίστης και στην ελευθερία της μη πίστης. Γιατί υπάρχουν πολλά άτομα ανά τον κόσμο, θύματα διακρίσεων, για να μην πω κάτι χειρότερο, μόνο και μόνο επειδή εκφράζουν τη δική τους ελεύθερη σκέψη, η οποία λέει συνοπτικά ότι δεν πιστεύουν σε κανένα Θεό. Πρέπει να υπερασπιστούμε και τους μεν και τους δε. Για την τρομοκρατία. Δεν συμφωνώ με την προσέγγισή σας απόλυτα. Νομίζω ότι η καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας δημιούργησε πολλέ καταχρήσει. καταχρήσεις. Λίγο-λίγο λέγεται αυτό. Γιατί το δικαίωμα στην ασφάλεια, το οποίο είναι θεμελιώδε βέβαια, επέτρεψε να προχωρήσουν κάποια πράγματα, τα οποία όμω, όποιο και είναι το πλαίσιο, δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Να υπερασπιστούμε, το να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σημαίνει να τα προωθούμε κάθε στιγμή και να μην ε, προωθούμε τη μία το ένα, την άλλη το άλλο. Κάθε φορά να έχουμε αυτό το μέλημα πρώτο, τα, ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση, η χρηματοπιστωτική κρίση βαραίνει κάποια πράγματα, λέτε, αλλά δεν, δεν μου αρέσει ο τρόπος που το λέτε. Π.χ. κάτι που αφορά την ε, Ευρώπη. Στο Ενωμένο Βασίλειο, εκατομμύρια στερλινών εγκα... δαπανήθηκαν για να εγκατασταθούν παντού βιντεοκάμερες σε όλη την επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι εργαλείο κατά πολέμης τρομοκρατίας, οι κάμερες. Ε, καθησυχάζει τους πολίτες, μερικές φορές βρίσκουμε και κάποιους ενόχους, αλλά δεν δημιουργεί πραγματική ελευθερία, πραγματική ασφάλεια στους πολίτες. Ίσως θα μπορούσαμε, ε, χρησιμοποιώντας καλύτερα τα λεφτά αυτά, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να προστατεύουμε παράλληλα και τους πολίτες. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρουμε την συνέπεια των μεταναστευτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα βάλουμε και τάξη και στον οίκο μας. Δεν μπορούμε να στέλνουμε πίσω, ας πούμε, μετανάστες στη Λιβύη, Φερρυπίνα, αλλά και αλλού, χωρίς να ανησυχούμε εμείς στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί θα του συμβεί μετά. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο. Και νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Κάποια μικρά σημεία για το Ιράν. Μιλάτε για τους ε, εγκληματίες ανηλίκους. Μην τους λέτε εγκληματίες. Είναι, υπάρχουν ανήλικοι που καταδικάζονται. Ένας 16χρονος ας πούμε που καταδικάζεται για σοδομισμό, για μοφιλοφιλία. Ε, δεν είναι εγκληματίας παρότι καταδικάζεται. Ε, Πρέπει να το καταδικάσουμε αυτό. Ε, τώρα, το βραβείο Σαχάροφ. Ε, πολύ ενδιαφέρον πέρυσι. Ένας από τους βραβευθέντες φυλακίστε, φυλακίστηκε αμέσως μετά το βραβείο αυτό. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έκανε ό,τι θα μπορούσε να είχε κάνει για να αναγκάσει στην απελευθέρωσή του. Επίσης, Πρέπει να δώσουμε σημασία στη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, όπως το λέτε ακριβώς. Συμφωνώ. Ε, από την άλλη όμως θα πρέπει να δώσουμε ίση ε, σημασία στη συνεργασία με τον ΟΗΕ. Αυτά και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι μακρηγορήσατε πολύ περισσότερο από τους άλλους συναδέλφους. Απλώς αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα γιατί πρέπει να δώσουμε το λόγο στους φίλους μας από τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά θέλω να δώσω το λόγο και στην κυρία Χιμένεθ και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο τέλος στην εισηγήτρια. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη κυρία Πρόεδρε γιατί ξέρω ότι έχουμε λίγο χρόνο. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια για την λαμπρότητα της έκθεσής της που έχει μια πολύ θετική προσέγγιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κριτικό πνεύμα κυρίως όμως προσπαθεί να κάνει επικοδομητική κριτική. Αυτός είναι και ο στόχος ύπαρξής μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κόσμο όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι απλώς φραστικό σχήμα αλλά πραγματικότητα. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα την κυρία Αντρίκενε για το κεφάλαιο που αφορά τη βία κατά των γυναικών. Πιστεύω ότι έχει διατυπωθεί πολύ σωστά. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κατάσταση πολλών γυναικών στην Ευρώπη που λόγω πολιτιστικών ή θρησκευτικών λόγων ζουν σε ένα είδος δουλείας από τις οποίες πολύ σπάνια μπορούν να βγουν. Έχουμε τα παραδείγματα των νέων κοριτσιών στις χώρες μας που πολλές φορές δολοφονούνται γιατί θέλουν να ζήσουν μια διαφορετική ζωή. Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών και για να μπορέσουν να βγουν από τον ασφυκτικό οικογενειακό κλειό όπου πολλές φορές ζουν σε κατάσταση δουλείας. Ένα άλλο κεφάλαιο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το κεφάλαιο που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Θέλω να συγχαρώ την κυρία εισηγήτρια για το γεγονός ότι περιλαμβάνει και αυτό το σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να μας επηρεάσει τόσο πολύ. Όταν αντιμετωπίζουμε το θέμα της τρομοκρατίας σε συνδυασμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό <clears throat> γίνεται πολλές φορές βλέποντας μονάχα την οπτική γωνία του επιτιθέμενου, του τρομοκράτη και μόνο. Σχεδόν ποτέ δεν αναφέρεται το, η κατάσταση των θυμάτων. Είναι απαραίτητο όταν μιλάμε για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας να λάβουμε υπόψη και τα δικαιώματα των θυμάτων που πολλές φορές χάνουν και τη ζωή τους ακόμα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτό τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τα θύματα της τρομοκρατίας και επομένω είναι απαραίτητο να αναφερθεί και στην έκθεση τη κυρία Αντρέκερα. Είναι απαραίτητο επίση να καταγγείλουμε τι κυβερνήσει που συνεργάζονται με, τον διεθνή, με τη διεθνή τρομοκρατία και που διώκουν την τρομοκρατία στο έδαφο του ακόμα και τον χρηματοδοτούν. Αυτό το βλέπουμε με πολλέ περιπτώσει απαγωγών που έχουν γίνει. Και επίση, σε ό,τι αφορά την Κούβα, μου φαίνεται ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να αναφερθεί το γεγονός ότι πολλοί από τους πολιτικούς κρατουμένους έχουν εκδιωχθεί από την Κούβα, δεν είναι πια στις αλλά έχουν εκδιωχθεί και δεν μπορούν να επανέλθουν. Πρέπει να επιμείνουμε λοιπόν για να υπάρξει ελευθερία όλων των κρατουμένων συνείδησης και στη χώρα αυτή και σε άλλες χώρες. Και σας συγχαίρω και πάλι κυρία να Ευχαριστώ πολύ κυρία Χιμένες. Ο κύριος Τίμονς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύντομα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Καταρχά θα ήθελα επίσης εξ ονόματο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγχαρώ την κυρία Αντρική Ένε για την πάρα πολύ καλά δομημένη έκθεση αλλά και την τόσο περιεκτική και συνολική. Το είπε και ο κύριος Χάουιτ. Εδώ και πολλά χρόνια το Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί τις εκθέσεις αυτές για να ασκήσει τον έλεγχό του και να λογοδοτούν στο Κοινοβούλιο τα άλλα θεσμικά όργανα για το τι πράττουν ή τι δεν πράττουν ε, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι σε τρίτες χώρες. Ε, ε, Μερικά σχόλια μου επιτρέπετε μόνο να κάνω για ορισμένα σημεία. Στην παράγραφο 12 που γίνεται λόγος για τις πολιτικές και τις προτεραιότητες αναχώρα. Θα ήθελα απλώς να σας ε, θυμίσω ότι προς αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε. Η αντίστοιχη ομάδα εργασίας του Συμβουλίου θα εξετάσει ένα προσχέδιο και πώς στο μέλλον θα γίνονται εκθέσεις αναχώρα. στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάντα. Και από την επόμενη χρονιά θα αρχίσουμε με ορισμένε πιλωτικέ χώρε για να τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 13 ε, και τους ενδεικτικούς δείκτες και σχετική αξιολόγηση και ορόσημα, ποιος το είπε αυτό, ο κύριος Χάουιτ επίσης και εκφράζει παράπονα ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα δεν έχουν ορίσει ε, σημεία παραμέτρους για συγκριτική αξιολόγηση και μέτρηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας των δράσεών μας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να πω ότι ε, γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να θέσουμε εκεί δείκτες και ορόσημα συγκρίσιμα. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό τον καιρό κάνει μια ευρύτατη ε, αξιολόγηση των πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων ε, δικαιώματα συγγνώμη, συμπεριλαμβανομένων και των ε, διαφόρων μέσων που έχουμε και των οικονομικών και θα ολοκληρωθεί περίπου ε, τα μέσα του θέρους του 2011. Θα είναι τότε λοιπόν μια καλή ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα τη συγκριτική αξιολόγηση και των δικτών και των ορισμών. Για το 54 θέλω να πω ότι κατά την άποψή μας Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι εννοεί η παράγραφος. Να εγκαθιδρυθεί ένας διοργανικός μηχανισμός συνεργασίας για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι θα πει αυτό και άλλος μηχανισμός για να αξιολογεί τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των καθευθυντήριων γραμμών. Αν μου επιτρέπετε, θα πρότεινα να αναδιατυπωθεί αυτή η παράγραφος, να γίνει πιο σαφής για το τι ακριβώς επιθυμείτε. Και στην ίδια παράγραφο επίσης θα πρόσθετα και κάτι ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, θα πρέπει, έχει δημιουργήσει θέσεις ε, που παρακολουθούν και ασχολούνται εξωτερικές αντιπροσωπίες ας πούμε σε αποστολές ε, των κρατών μελών όπου έχει κατανεμηθεί και η αρμοδιότητα όχι στο εσωτερικό όμως των θεσμικών οργάνων. Η παράγραφος 59. Μία εκτίμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα για χώρες τρίτες με τις οποίες συνάπτουμε συμφωνίες. Τι εννοείται κυρία Αντρικέρη, μια επέκταση ε, των ε, μελετών ε, δικτύπου και επιπτώσεων σε εμπορικές συμφωνίες αυτή τη στιγμή περιορίζονται μόνο στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κτλ. Αυτό ζητάτε. Γίνεται αυτή η συζήτηση, αλλά νομίζω ότι και αυτό χωράει διευκρίνηση. Στη συνέχεια, στο σημείο 76, κατανοώ ότι μπορεί να διαφέρουν οι θεωρήσεις και απόψεις ε, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής από αυτού, αλλά και του Συμβουλίου. Γίνεται λόγος για έλλειψη προόδου ε, στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διαβουλεύσεις. Κοιτάξτε, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε οι διαπραγματεύσει αυτέ και οι διαβουλεύσει και ο διάλογο να έχουν πρόθεσμε επιπτώσει και αποτελέσματα. Αυτό είναι μακρά πνοή. Μέσω πρόθεσμα, μακροπρόθεσμα θα πρέπει να κάνουμε τι χώρε να αλλάξουν στάσει και συμπεριφορέ. Ε, ισχυρίζομαι ότι έχουμε και πρόοδου και επιτυχίε αυτό. Αν θέλετε να το συζητήσουμε άλλη ώρα σε λεπτομέρειες. Αλλά βέβαια είναι ε, εξουσία του Κοινοβουλίου αυτό. Αλλά εγώ θα μιλούσα γενικά για απογοήτευση. Συγγνώμη, διακόπτη πρόεδρος, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Ναι, για την κοινωνία των πολιτών θα θυμίσω ότι έχουμε σεμινάρια για τους πολίτες, τακτικά κιόλας. Βέβαια όχι συστηματικά, αλλά πάρα πολύ συχνά είναι και θέμα αρχή πάντα στι τρίτε χώρες. Τελευταία παρατήρηση. λέσαν πολλοί συνάδελφοι ε, την εκπαίδευση, κατάρτιση προσωπικού. Εκατοντάδε υπαλλήλου εκπαιδεύσαμε τα τελευταία χρόνια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρει-τέσσερι φορέ το χρόνο ειδικά μαθήματα. Αλλά στο μέλλον θα καταρτίζουμε και θα επιμορφώνουμε καλύτερα συγκεκριμένα και στοχευμένα τις αντιπροσωπείες που θα πηγαίνουν στις διάφορες χώρες. Αυτά. Και πάλι θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Αντρική Ενέ για την εξωτερική έκθεσή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι σίγουρο, σίγουρη ότι η συγγήτρια έχει κατανοήσει ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο έχει διαθώσει την έκθεσή της και έχει καταγράψει πιστεύω τις κύριες μέρημνες των βουλευτών που ζητούν μια μεγαλύτερη ισορροπία παρά το γεγονό ότι φυσικά δεν πρέπει να κατανομάζονται συγκεκριμένε χώρε. Ο κύριο Πρόντι και η κυρία Νίτσεν αναφέρθηκαν ορισμένα ζητήματα που συνάπτονται με το περιβάλλον. Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο και η ίδια η συγγήτρια τόνισε για την κλιματική αλλαγή. <coughs> Μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε μερικά τέτοια θέματα το θέμα των μειονοτήτων, το θέμα τη διεθνού ποινική δικαιοσύνη αναφέρθηκε, η ανάγκη να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και επίση να δούμε το πώ το Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει μια άποψη για την έκθεση Goldstone και αυτό θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη. Το θέμα τη μετανάστευση ω πολιτική όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει απόλυτα τις υπόσχεσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με όλα αυτά θέλω να ξαναδώσω το λόγο στην κυρία εισηγήτρια και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για καλύτερα, ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ λέει, κύριε Αντρικάινε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω πρώτα απ' όλα ότι πρόκειψε μια τεράστια σύγχυση. Όλα τα σημειώματά μου, όλες οι σημειώσεις μου ήταν στα λιθουανικά και αναγκάστηκα να μιλήσω αγγλικά. Περίμενα τουλάχιστον σήμερα να υπάρχει διερμηνία στα... από τα λιθουανικά. Σας ζητώ συγγνώμη λοιπόν για το γεγονός ότι μπορεί να μην στάθηκα ιδιαίτερα σαφής στην αρχή όταν έλαβα το λόγο. Απαντώντας τώρα σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας και για τις παρατηρήσεις σας. Κατέγραψα όλα αυτά τα οποία είπατε Ρίτσαρντ ε, Χάουιτ. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Αλλά επειδή είμαι μέλος αυτής της υποεπιτροπής εδώ πολύ καιρό, καταλαβαίνω ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σύστημα GSC, η ελευθερία της ε, ε, θρησκευτικής πίσης, μετανάστευση, επιπτώσεις χρηματοοικονομικής κρίσης, τρομοκρατία, όλα αυτά τα οποία ανέφερες, τα, θύματα, τα δικαιώματα των θυμάτων της τρομοκρατίας, το θέμα της ε, βίας κατά των γυναικών, η πίεση στους φυσικούς πόρους, όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι τα έχω υπόψη μου και θα προσπαθήσουμε να βρούμε ίσως μια καλύτερη συμβαστική ε, κοινή θέση στην έκθεση. Εγώ έχω υποσχεθεί ότι θα προσπαθώ να είμαι όσο δυνατόν πιο περιεκτική. Είναι προφανώ δική μου έκθεση, αλλά είναι και η έκθεση που θα αποτελέσει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι το ψήφισμα λοιπόν και η έκθεση όλων μα. Έτσι κατανοώ τα πράγματα. Ελπίζω λοιπόν επίσης ότι η πρόεδρος θα προτείνει και κάποιο, κάποια προθεσμία πιο ευρεία για την κατάθεση τροπολογιών. Κάτι ακόμα. Έχουμε και την Στογγυλή Τράπεζα την επόμενη εβδομάδα στις 3 η ώρα, στη 1.30, μια Στογγυλή Τράπεζα με τους μη κυβερνητικού φορείς για τα αισθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί από εσάς λοιπόν που ενδιαφέρονται να ακούσουν τις απόψεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είσαστε παραπάνω από καλόδεκτοι την Τρίτη στη μία μισή, την επόμενη Τρίτη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχόλια τα οποία μας έδωσε. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστούμε πολύ κυρία εισηγήτρια. Οι υπηρεσίε μας έχουν συζητήσει για την, το θέμα των προθεσμιών που δεν είναι ικανοποιητικές για σας. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μία μείζωνα συζήτηση για αυτό το θέμα και άλλα θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το ραντεβού. Θέλω όμως να υπάρχει διαφάνεια. Χρειάστηκε πολλοί στις πολιτικές ομάδες για να καθορίσουν ποιος θα είναι εισηγητής. Χάσαμε την αρχή της διαδικασίας. Μπορούμε τώρα να παρατείνουμε την ε, προθεσμία της τροπολογίας κατά μία εβδομάδα, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Αν δέχεστε οι τροπολογίες να κατατεθούν μόνο στα αγγλικά ή στα γαλλικά, μπορούμε να παρατείνουμε την προθεσμία των τροπολογιών μέχρι το μεσημέρι της 14ης Οκτωβρίου. Δηλαδή μια εβδομάδα παραπάνω. Δεν μεχρι το μεσημερι της 14 η οκτωβριου δηλαδη μια καλύτερη πρόταση να σας κάνω λοιπόν. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να παραμείνουμε στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που μας φέρνει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. How it. Αν μπορώ να βοηθήσω λιγάκι για τις άλλες γλωσσικές κοινότητες. Υποθέτω ότι αν υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θέλουν να καταθέσουν τις ε, τροπολογίες στη δική τους γλώσσα μέχρι την επόμενη Παρασκευή, ότι αυτό θα μπορούν να το κάνουν ούτως ή άλλως νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ του βουλευτέ μας που δεν θέλουν να καταθέσουν τροπολογίες στα αγγλικά και γαλλικά. Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτή θα είναι μια πολύ καλή συμβαστική λύση για αυτή την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν άλλε γλώσσε τη τροπολογία θα πρέπει να παραμείνουν στο αρχικό πλαίσιο, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι τη 7η Οκτωβρίου, αλλά αγγλικά-γαλλικά στι 14. Εγώ διαμαρτύρομαι, λέει κυρία Βεζιά, αυτά είναι εγώ Μεγαλίδα, αλλά αυτό με βολεύει. Αλλά δεν μπορούν όλοι οι βουλευτές να μην έχουν τις ίδιες συνθήκες εργασίας. Αυτό δεν είναι παραδεκτό. Είναι ένα σκάνδαλο αυτό για μένα. Η μόνη πρόταση που μπορώ να σας κάνω, λέει η Πρόεδρος, είναι ότι θα φέρω το θέμα αυτό στην συνέλευση του διευρυμένου μας Προεδρείου το μεσημέρι στις 2 και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω μια καλύτερη πρόταση και νομίζω ότι και ο κύριος Χάουιτ έχει λάβει υπόψη την κατάσταση των υπηρεσιών. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο διευρυμένο προεδρείο της Επιτροπής μας. Και τώρα μου είπανε ότι επειδή έχουμε τη συνάντηση αυτή στις 2 η ώρα, οι διερμηνείς πρέπει να σταματήσουν στις, στις 12.30. Καταλαβαίνω ότι έχουν δικαίωμα διακοπής. Πρέπει λοιπόν να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί αντί για μία ώρα για να συζητήσουμε την πρωτοβουλία ΡΕΚΟΜ που είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της βάσης που θέλει να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έχουμε μονάχα μισή ώρα. Ε, αλλά συζητήσαμε την πιο σημαντική έκθεση του χρόνου και ελπίζω ότι όλοι οι ομιλητέ θα μπορέσουν να προσαρμόσουν το χρόνο παρέμβασή του για να μην μειώσουμε τον αριθμό των ομιλητών. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Κούκαν που είναι μέλο τη υποεπιτροπής μα, ο οποίο μα έφερε σε γνώση μα την πρωτοβουλία Ρέκομ και τα, τους στόχους της. Η ΡΕΚΟΜ είναι η Περιφερειακή Επιτροπή για την Αναζήτηση και την Αποκάλυψη της Αλήθειας σε σχέση με τα εγκλήματα που έχουν λάβει η χώρα στην πρώην Ιουκοσλαβία. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πιέρ Μιρέλ, ο οποίος είναι ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Διεύθυνσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επαφές που είχε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δοθεί αυτή η δυνατότητα να ενισχυθεί αυτή η σημαντική πρωτοβουλία. Το πλαίσιο λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι ο πόλεμος στην πρώην Ιουκοσλαβία οδήγησε σε εκατοντάδες ε, χιλιάδες ουσιαστικά θανάτων και πάνω από δύο εκατομμύρια εκτοπισμένων. Υπάρχουν πολλά άτομα που είναι ακόμα αγνοούμενοι, κάτι που αποτελεί μια τεράστια τραγωδία για τους οικείους τους. Υπάρχουν ε, μαζικοί τάφοι που δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί και υπάρχουν υποψίες για μαζικά εγκλήματα πολέμου. Το παράδειγμα τη γενοκτονίας τη Ρεμπρένιτσα είναι μόνο ένα παράδειγμα από τα εκκρεμή θέματα τα οποία δεν έχουν διαλευκανθεί. Το ζήτημα είναι αν οι πολιτικέ ελίτ τη χώρε αυτέ που προέκυψαν τη διάλυση τη Ιουγκοσλαβίας κάνουν μια ουσιαστική προσπάθεια συμφιλίωσης. Θέλουμε να δώσουμε μια μεγάλη ορατότητα σε αυτή την πρωτοβουλία τη βάση τη ΡΕΚΟΜ η οποία έχει προσκληθεί εδώ από τον κύριο Κούκαν ο οποίος είναι Μέλο τη αντιπροσωπεία για τη σχέση με τι χώρες της Νοτιοανατολική Ευρώπη και ο οποίο θα διευθύνει αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Θα σα ευχαριστήσω λοιπόν για την παρουσία σα Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κούκαν. Έχουμε πολλού καλεσμένου οι οποίοι συμμετέχουν στην στρογγυλή τράπεζα αυτή η οποία κανονικά λαμβάνει χώρα εκτό τη συνεδριασής τη Επιτροπής μας. Και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κούκαν για να προεδρεύσει αυτή την ημίωρη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι και δική μου χαρά που καλωσορίζω τους διακεκριμένους καλεσμένους της πρωτοβουλίας RECOM. Λόγω του περιορισμένου χρόνου θα είμαι πολύ σύντομος στις παρατηρήσεις μου, ούτως ώστε να τους δώσω περισσότερο χρόνο. Καταρχάς, Σας καλωσορίζω θερμά και ειλικρινά. Όπως βλέπετε κι εσείς, ο δρόμος προς τις Βρυξέλλες δεν είναι καθόλου εύκολος. Ο πολιτικός αυτός δρόμος δεν είναι καθόλου εύκολος. Αλλά και φυσικός πώς δεν είναι εύκολο να φτάσει κανείς στις Βρυξέλλες. Λόγω της απεργίας, της μεταφορές, ε, δυσκολευτήκατε να, βρείτε τον να φτάσετε στον προορισμό σας, στις Βρυξέλλες. Σας καλωσορίζω λοιπόν και όπως βλέπετε αντί για μία ώρα σας δίνουμε μόνο 30 λεπτά. Η ζωή στις Βρυξέλλες είναι πολύ δύσκολη τελικά. Η κυρία Πρόεδρος είπε ε, ποια, είναι, τα βασικά θέματα της ε, πρωτοβουλίας αυτής. Ποια είναι η ατζέντα που έχουμε στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας. Ε, με αυτά τα κύρια θέματα που ανέφερε η Πρόεδρος περιγράφεται και αυτή η πρωτοβουλία πολύ σωστά. Θέλω να τονίσω ότι η πρωτοβουλία αυτή ε, εκφράζει επαρκή, επαρκώς όλες τις χώρες. Υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα σωστή από όλες τις χώρες της περιοχής και αυτό δείχνει την θέληση των χωρών να συνεργαστούν για αυτά τα πολύ ευαίσθητα θέματα. Επίσης, Είναι πολύ σημαντικό, σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και σε διεθνές πλαίσιο. Μην, μιλάμε για, μην ξεχνάμε για μια άλλη πρωτοβουλία που είναι το εφαλτήριο για τη διαδικασία ε, συμφιλίωσης. είναι η ενδιάμεση αυτή, μεταβατική αυτή δικαιοσύνη. Ε, αυτή η διαδικασία ε, είναι κατ' εικόνα και ομοίωση της διαδικασίας που έλαβε χώρα και στη Νότια Αφρική. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ζητάμε ε, τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής με συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το τη συζήτηση εδώ σήμερα. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες συζητήσεις και άλλα φόρουμ. Αυτή η πρωτοβουλία φυσικά έχει μια περιφερειακή σημασία. Η φύση των εγκλημάτων ήταν περιφερειακή και επομένως αφορούσε την περιοχή αυτή. Ε, αφορούσε όλη την περιοχή και επομένως δεν είχε νόημα να αντιμετωπίσουμε τα εγκλήματα αυτά κατακαιρματισμένα σε κάθε χώρα. Κάτι άλλο ο, εντοπισμός, των εγκληματιών, ούτω ώστε να παρεμποδίσουμε μια γενικευμένη κατάσταση εγκλήματος και να μην υπάρξουν γενικώ κατηγορίες προς δικαίους και αδίκους. Και αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Συνοψίζω, η ΡΕΚΟΜ είναι η πρωτοβουλία αυτή που αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια όπου δραστηριοποιούνται πολλά άτομα ε, με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ήταν μια εισαγωγή. Τώρα θα δώσω το λόγο στους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας. Σας παρακαλώ καταλάβετε μας και προσπαθήστε να είστε ως τον πιο λακωνικοί. Μπορείτε να μιλήσετε για δύο λεπτά. Δυστυχώς, αν ξεπεράσετε αυτό το χρονικό όριο, θα είμαι σκληρός. Θα χρησιμοποιήσω το σφυράκι μου, θα σας το πετάξω. Αλλά απλώ να σας δείξω ότι τέλειωσε ο χρόνος σας. Η κυρία Νατάσα Κάντιτς από τη Σερβία, από το Κέντρο Ανθρωπιστικού Δικαίου. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Χαουτάλ, ευχαριστώ κύριε Χούκαν, Κούκαν και σας κύριε Μιρέλ. Σας ευχαριστώ για αυτή τη θαυμάσια πρωτοβουλία που μας δίνετε και να παρουσιάσουμε την πρωτοβουλία μας που ονομάζεται RECOM. Είναι μια τοπική απάντηση στις τοπικές ανάγκες που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το παρελθόν μας. Είναι μια απόπειρα να απαντήσουμε στα όσα λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ιουγκοσλαβία με ανοιχτά τα μάτια και να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Ξέρουμε ότι οι δίκες αφορούσαν, που έχουν γίνει μέχρι στιγμής αφορούσαν τους εγκληματίες όσους διέπραξαν αδικήματα. Στις δίκες, ειδικά στις εθνικές δίκες, υπάρχει μία πολιτική και μία εθνική διάσταση πάντα. Με το ρέκο. όμως θέλουμε να ξεπεράσουμε τους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς περιορισμούς των δικών. Θέλουμε να αναπτύξουμε αλληλεγγύη στις κοινωνίες μας και συμπόνια απέναντι σε όλα τα θύματα. Οι συνάδελφοί μου θα μιλήσουν περισσότερο για την υποστήριξη που έχουμε με αυτή την πρωτοβουλία. Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε την αφοσίωσή μας Προ μια προσπάθεια δημιουργία ενός περιφερειακού φορέα που θα ασχοληθεί με τα θύματα, όχι με τους ε, διώκτες και τους εγκληματίες. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη θαυμάσια ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την προσπάθεια. Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και για το γεγονό ότι καταλαβαίνετε ποια είναι τα χρονικά όρια. Η κυρία Βέσνα Τέρσελιτ από την οργάνωση Documenta, Κροατία. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω, μας ενθαρρύνει πάρα πολύ η υποστήριξη ε, του κυρίου Πιρέλ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι τώρα και ελπίζω να εξακολουθούν να μας υποστηρίζουν και στο μέλλον. Και μέχρι τώρα είναι εξαιρετική υποστήριξη. Έχουμε πάνω από 900 οργανώσεις ε, μεμονωμένες οι οποίες συμμετέχουν στη δική μας πρωτοβουλία ενός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης ε, από τις ενώσεις αγνοουμένων, ε, κρατουμένων, εκτοπισμένων, γυναικείων οργανώσεων, πολεμάχων και διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων και πιστών. Επίση, έχουμε δεχτεί υποστήριξη του Προέδρου τη Κροατία, του κυρίου Γιωσίποβιτ και του Πρόεδρου ε, Τάντιτ της Σερβίας. Τώρα συζητούμε με διάφορα ε, κόμματα και κυβερνητικές οργανώσεις και θεσμούς γιατί είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη συγκυρία. Ε, προωθούμε την εκστρατεία μας και ε, στο Ζάγκρεμπ και στο Σαράγεβο. Και τώρα περιμένουμε και την υποστήριξη των κοινοβουλίων των χωρών μας. Και του χρόνου θα υποβάλουμε τις προτάσεις στα κοινοβούλια στους προέδρους των κρατών για να συσταθεί αυτή η Επιτροπή. Από το 2006 γίνεται λόγος για αυτό, αλλά μόνο οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια ε, μπορούν να συμφωνήσουν για να τεθεί σε ισχύ. Ε, γίνεται λόγος ε, για το καθεστώς, για το καταστατικό που θα ορίζει ποιος θα είναι μέλος ε, ποια θα είναι οργανωτική, οργανωτική δομή. Ε, έχουμε μικρές συνεδριάσεις μεταξύ 30 και 70 ε, μελών και μέχρι και 200 μέλη έρχονται στις συγκεντρώσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Τζινάνα Καροτρούσκο από την Ένωση δημοσιογράφων Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ευχαριστώ πολύ. Το ποινικό δικαστήριο νομίζω ότι έχει κάνει ένα μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας. Στη Βοσνία Ζεγοβίνη υπήρξαν τόσα πολλά εγκλήματα πολέμου που τα δικαστήρια δεν έχουν την ηλική δυνατότητα να διεκπαιρεώσουν όλες τις μεμονωμένες υποθέσεις και να καταλήξουν στο τι ακριβώς έγινε μπορούν να έχουν μονάχα την λεγόμενη δικαστική αλήθεια. Εμεί χρειαζόμαστε όμω μια πιο πλήρη διαδικασία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα του παρελθόντος. Μόνο όταν γίνει αυτό θα μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση. Η Βοσνία Ζεχοβίνης δεν μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να έχουμε και τα απαραίτητα στοιχεία από το Βελιγράδι ή από το Ζάγρεπ. Γιατί ό,τι έγινε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας χρειάζεται και την αρρωγή των χωρών αυτών. Τον Οκτώβριο θα γίνουν εκλογές στη Βοσνία Ερσεγοβίνη και μετά από αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε την αλήθεια. Υπάρχει ακόμα η άρνηση των εγκλημάτων αυτών που έχουν γίνει. Ο πρόεδρος της Ρεπούμπλικα Σρεψκα είπε ότι δεν υπήρξε καμία γενοκτονία στην ε, Σρεμπένισσα. Θα χρειαστούμε λοιπόν μεγάλη δύναμη για να έχουμε υποστήριξη όλων των πλευρών για την αλήθεια στην περιοχή αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριο Κούκαν. Ο κύριο Σούμπιν Μουσίτ από την Ένωση των Κρατωμένων ε, πριν από το 1992 στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Μούσιτ λέγομαι και θα λάβω το λόγο σε σχέση με την, την οργάνωση Πρίατορ 1992 που αφορά τους ε, επιβιώσαντες από τα χειρότερα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στον κόσμο μετά από το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στην πρωτοβουλία και την ανάγκη που υπάρχει. Απλώς θέλω να σας πω σε ποιο βαθμό η κοινωνία της Βοσνίας Ερζεχοβίνης έχει αντιμετωπίσει το παρελθόν για τα θέματα αυτά. Αντιμετωπίσαμε ένα ολοκαύτωμα, ένα εργοστάσιο θανατώσεως. Μια εταιρεία ευρωπαϊκή δημιούργησε αυτό το στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Πάνω από 200 άτομα σκοτώθηκαν εκεί σε αυτό το στρατόπεδο μέσα σε ένα βράδυ. Και τώρα χρησιμοποιείται για τη βαφή αυτοκινήτων. Στο τέρμα Πόλια υπήρξε ένα στρατόπεδο στο οποίο έχουν ε, βρεθεί για το στρατόπεδο αυτό φωτογραφίες κρατουμένων που πέθαναν γιατί τους εξανάγκασαν σε λοιμό, σε έλλειψη τροφίμων. Όλα αυτά λοιπόν αυτα, λοιπον ακομα δεν έχουν διαλευκανθεί στην ε, Βοσνία Ζεχοβίν. Εγώ έχω περάσει και ο ίδιος ως ανήλικος από στρατόπεδα συγκεντρώσεων. Κάποια άτομα λοιπόν επανέρχονται και στη χώρα μου και βλέπω ότι τίποτα δεν γίνεται στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Απλώς έχει συντελεστεί εθνοτική κάθαρση. Υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη να υπάρξει μια περιφερειακή δράση για να αντιμετωπίσουμε το παρελθόν. Όσο δυνηρό και να είναι το παρελθόν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αν θέλετε η Βοσνία Ζεγοβίνη να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κούκαν, δεν θέλετε να υπάρχουν μεγαλύτερες διαδηλώσεις μέχρι να καταλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μας ε, υποστηρίξει. Ευχαριστώ. Τάλι Μπόρκα Ουλιαρέβιτς από το κέντρο ε, πολιτικής εκπαίδευσης στο, Μαυροβούνιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δική μας πρωτοβουλία, για την υποστήριξή σας. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε έτσι τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει μέχρι τούδε και μας ενθαρρύνετε για να συνεχίσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιόν μας. Είναι μια πολύ σύνθετη αυτή η πρωτοβουλία με πολλές προκλήσεις, αλλά ήδη έχουμε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για την περίπτωση του Μαυροβουνίου. Εμείς δεν είχαμε εδώ και δύο δεκαετίες θέση στην ατζέντα μας ε, το θέμα του παρελθόντος πριν ξεκινήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Με αυτό τον τρόπο δείχνουμε ότι μόνο περιφερειακά αν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από την άλλη, έχουμε και την υποστήριξη του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου. Όλες οι πολιτικές, τα πολιτικά κόμματα και ομάδες έχουν υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντική για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ελπίζω με τη δική σας υποστήριξη θα υπάρξει πολιτική υποστήριξη και στις υπόλοιπες χώρες για την πρωτοβουλία ΡΕΚΟΜ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Δράγκαν Πιέβατς από την Οργάνωση Οικογενειών των αγνοούμενων και Δολοφονημένων από την Κραίνα της Σερβίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε το χρόνο να μιλήσουμε και είστε διατεθειμένοι να μας ακούσετε για αυτά τα πολύ δύσκολα θέματα. Θα πω κάποια πράγματα από τη σκοπιά του θύματος. Ακόμα και τα θύματα υποστηρίζουν την πρωτοβουλία ΡΕΚΟΜ και τη θεωρούμε πραγματικά εκ κάνευ. Η μητέρα μου δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο στα 66 της. Αυτή λοιπόν μου έλεγε ότι κουφός είναι αυτός που αρνείται να ακούσει. Τα κόμματα στη Σερβία και στην Κροατία δεν μπορούν να ακούσουν για αυτά τα θέματα. Δυσκολεύονται και αν το κάνουν, μόνο προτάσουν τα δικά τους θύματα και παριστάνουν οι ίδιοι τα θύματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την υπομονή σας σήμερα. Δεν είναι τυχαίο που μια τέτοια πρωτοβουλία είναι σε θέση να προκαλέσει αυτές τις συζητήσεις. Σας ευχαριστώ και πριν, από, πριν έρθω σήμερα εδώ είχα πάει και στο Κοινοβούλιο της Κροατίας και της Σερβίας. Σας ευχαριστώ και τώρα η κυρία Σβετλάνα Βούκοβιτ στο Κέντρο για την Υπεύθυνη Δημοκρατία. Λούνα Ρούντο, Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σα ευχαριστήσω. για την ευκαιρία που μας έχετε δώσει να παρουσιάσουμε την πρωτοβουλία μας ενώπιόν σα. Η Ένωσή μου είναι μέλος της ε, σύμπραξης της Συμμαχίας ΡΕΚΟΜ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στο να υπάρξει μια περιφερειακή επιτροπή στα Βαλκάνια, στην Προγικοσλαβία, για να διακριβώσει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι γεγονός ότι στα τελευταία 15 χρόνια οι περισσότερες από τις χώρες μας αντιμετωπίσανε στενά εθνοτικές προσεγγίσεις και χρειάζεται να υπάρχει η θέληση σε μια Περιφερειακή Επιτροπή να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό με τρόπο ολοκληρωμένο. Οι εθνικέ στρατηγικέ στην περιοχή δεν φτάνουν. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η περιφερειακή προσέγγιση για όλου μα στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Γκόρνταν Μπόσανατ, Κέντρο Ειρήνη και Δημοκρατία στην Κροατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά επιχειρήματα να παρουσιάζονται τα οποία δείχνουν γιατί είναι σημαντική η ΡΕΚΟΜ για τους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα να τονίσω τώρα τη σημασία της ΡΕΚΟΜ όχι μόνο για το λαό των Δυτικών Βαλκανίων αλλά για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η όλη διαδικασία της διεύνησης για τα Δυτικά Βαλκάνια έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Σύντομα αν όχι, αργότερα αν όχι σύντομα, οι χώρες αυτές οι οποίες έχουν περάσει μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία πολέμου θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την πολιτική διεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαδικασία σταθεροποίησης των Βαλκανίων. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αργά ή γρήγορα οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης <clears throat> θα έχουν μεταξύ τους τα θύματα των συγκρούσεων στα Βαλκάνια και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες αυτοί των Βαλκανίων να έχουν το καθεστώς των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με την προσχώρηση των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι μονάχα τα θύματα που θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες, αλλά και κάποιοι από τους δράστες των εγκλημάτων αυτών θα περιληφθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν θα έχουμε τον καιρό να τους διώξουμε όλους και να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Τέλος, η διαδικασία, η ιστορία της ε, σύγκρουσης στα Βαλκάνια δεν είναι μονάχα η εσωτερική ιστορία των χωρών αυτών, είναι και η ιστορία της σύνολης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με ένα εμπεριστατωμένο τρόπο για την ε, σύγκρουση αυτή στην πρώην είναι απαραίτητο να έχουμε τα πραγματικά γεγονότα στο μυαλό μας. Μόνο με δράσεις όπως η ΡΕΚΟΜ θα μπορέσουμε να γράψουμε πλήρως την εικόνα, την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να συμπεριλαμβάνει τα Βαλκάνια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν έρχεται αυτή η πρωτοβουλία στα κοινοβούλια των εμπλεκομένων χωρών, όταν αποκομίζει πολιτική υποστήριξη, να έχουμε κυρίως και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Τελευταίος, αλλά όχι ίστατος, Αυτήν Μερέντσαφ για, από την οργάνωση 22 Μαΐου Κόσοβα. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Έρχομαι από την οικογένεια Μελενίτσου από τη Βοστρία. Έρχομαι από μια χώρα που έχει μόλις εξέλθει από μια σύγκρουση που οδήγησε σε πλειάδα θυμάτων. Η χώρα μου έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές 22 Μαΐου είναι η ημερομηνία του 1999 όταν πολλοί από τους κατοίκους της πόλης μου σκοτώθηκαν ή έγιναν αγνοούμενοι. Είναι επομένως θύματα ενός πολέμου και εγώ ως επίσης θύμα αυτού του πολέμου ήθελα να πω γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη μια περιφερειακή πρωτοβουλία για τα θέματα αυτά και θα βοηθήσει και τα θύματα του πολέμου. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η πρωτοβουλία είναι γιατί πρέπει να βρούμε τους αγνοούμενους στις χώρες μας. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί έχουν δολοφονηθεί στο Κόσοβο και τα πτώματά τους ε, τα μπορεί να έχουν διασκορπιστεί σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε κάποια ακρίβεια σε σχέση με τα αριθμητικά στοιχεία που πολλοί χρησιμοποιούν αριθμούς οι οποίοι δεν είναι εδρεωμένοι στην πραγματικότητα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλα τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει στην περιοχή μας και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα να καταθέσουν αυτοί οι οποίοι έζησαν αυτά τα γεγονότα στο Κόσοβο να καταθέσουν την εμπειρία τους για όλα αυτά τα εγκλήματα. Θέλω και πάλι σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας και φυσικά η πρωτοβουλία αυτή αξίζει πιστεύω πλήρως την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους διακεκριμένους καλεσμένους μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι ήσασταν ιδιαίτερα λακωνικοί. Το μήνυμά σας ήταν ιδιαίτερα σαφές. Και θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Πιέρ Μιρέο, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο πατέρας αυτής της πρωτοβουλίας, ήταν παρόν τα ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και μπορώ να σας πω ότι και ο ίδιος ενεπλάκει με ιδιαίτερα ενεργό τρόπο για να εξασφαλίσει την επίσκεψή σας στις Βρυξέλλες. Δύο λεπτά πια, δύο λεπτά πια. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Ε, καθήκον μου το θεωρώ. Τρεις παρατηρήσεις πάρα πολύ σύντομα. Εγώ Πιστεύω ακράδαντα ότι η πρωτοβουλία ΡΕΚΟΜ είναι εκ των όν ως συμπλήρωμα προς το ε, δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου. Δεν νοείται συμφιλίωση, ούτε πρόκειται να επέλθει στα Δυτικά Βαλκάνια, χωρί αυτή την προσέγγιση από κάτω προ τα πάνω, που θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη υποστήριξη των κυβερνήσεων και των ε, κοινοβουλίων τη περιοχή. Η αλήθεια, η λογοδοσία και η συμφιλίωση θα πρέπει να προέλθουν ακριβώς από την ίδια την περιοχή αν θέλουμε να είναι διαρκής και βιώσιμη. Οι χώρες οι ίδιες θα πρέπει να ξεπεράσουν την κληρονομιά του παρελθόντος και οι προσπάθειες αυτές να γίνουν σε όλα τα επίπεδα, κυβερνητικό, δικαστικό, κοινωνία των πολιτών. Και γι' αυτό με τη δική μας υποστήριξη και την υποστήριξη ε, της πρωτοβουλίας ΡΕΚΟΜ πλήρως. Γι' αυτό και την υποστηρίζουμε και εμείς. Και η σημερινή ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τόσο σημαντική και θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς σας κυρία Πρόεδρε, προς την Επιτροπή σας και σας κύριε Κούκαν για την πλήρη υποστήριξη που δώσατε και εσείς στην προσπάθεια μας αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα αρχίζει η συζήτηση. Πρώτος ομιλητής, ο αξιόλογος ε, συνάδελφος Ζόραν Τάλερ, είναι Σλοβαίνος και πάρα πολύ δραστηριός και στην περιοχή αλλά και αλλού. Ευχαριστώ αγαπητέ ε, συνάδελφε κύριε Κούκαν. Ε, θα... Ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση προς όλους σας, τα σερβοκρότικα, ο κύριος Στάλερ. Χωρίς αυτή την προσπάθεια δεν πρόκειται να υπάρξει μέλλον και δεν πρόκειται να υπάρξει συμφιλίωση. Ε, γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα ε, ως προς τα πραγματικά περιστατικά και τα πραγματικά γεγονότα. Θα πρέπει να επηρεάσουμε σε όλες τις χώρες και τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης να βγάλουν την αλήθεια στην επιφάνεια. Πόσες γενιές θα χρειαστούν μέχρι να γραφτεί μια κοινή ιστορία αυτών των τόσο τρομερών φρικτών εποχών που ζήσαμε. Πόσες γενιές θα χρειαστούν για να είναι κοινά τα σχολικά χειρίδια για την περίοδο αυτή. Γνωρίζουμε ότι η Γαλλία και η Γερμανία το κατόρθωσαν μετά από φρικτούς πολέμους που τους χώριζαν και παγκοσμίους πολέμους. Οι Ιταλοί και οι Σλοβαίνοι είμαστε σε μια πρώτη φάση. Οι ιστορικοί ε, έγραψαν την κοινή ιστορία για ε, μια αιματοχυσία 100 ετών. Όχι λοιπόν μόνο στα Δυτικά Βαλκάνια και αλλού υπάρχει ανάγκη να επέλθει συμφιλίωση στην Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερο στα Ειδικά Βαλκάνια, να υποστηριχθούν τέτοιες πρωτοβουλίες για να έχετε και περισσότερο χώρο και περισσότερη ενέργεια και περισσότερα κονδύλια και περισσότερους πόρους. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ. υπόλοιποι συνάδελφοι για ένα λεπτό, κύριε Χιμένες. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς. Ευχαριστώ τους προσκαλεσμένους μας και κυρίως τον ε, τελευταίο μιλητή, τον κύριο Ντράγκαν. Ε, θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι δεν είμαστε κουφοί. Ότι, έχουμε, ότι, ακούμε και ανοίγουμε τα μάτια για την συμφιλίωση. Είναι πολύ σημαντικό. Μόνο στα πλαίσια της συμφιλίωσης μπορεί να υπάρξει αποζημίωση και στα θύματα, στήματα. Τα θύματα μόνο αυτό θα δεχθούν. Θα δεχθούν δηλαδή το προϊόν μιας διαδικασίας που θα οδεύει προς τη δικαιοσύνη. Βεργία. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω, όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές, τους φεχικλημένους μας και εσάς που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Και κρίμα που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Και εγώ θεωρώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, ότι η αποκατάσταση της αλήθειας είναι προϋπόθεση για να οικοδομηθεί το μέλλον. Μπράβο σας λοιπόν. Μπράβο για τη δουλειά σας. Μπράβο για το θάρρος σας. Εδώ στο Κοινοβούλιο είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι για αυτά τα θέματα και νομίζω ότι οι απόψεις μας συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό για αυτά τα θέματα. Θέλω να πω στους συναδέλφους ότι η Μεγαλίδα και η Γαλλία και η Γερμανία, πολύ περισσότερο μάλιστα η Γαλλία από τη Γερμανία, χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να χύσουν το φως στο παρελθόν τους. Και ακόμα υπάρχουν ε, σκοτεινές πτυχές για την ιστορία μας στη Γαλλία. Πολύ περισσότερο για τον πόλεμο στην Αλγερία παρά για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χρειάζεται χρόνος λοιπόν, αλλά δεν πρέπει να αποθαρρυνθούμε. Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Νομίζω ότι μόνο έτσι, μόνο με τις πρωτοβουλίες ε, θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε το μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, με περιορίζει ε, ο χρόνος. Ε, θα ήθελα να πω όπως και άλλοι συνάδελφοι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και σας ακούσαμε. Μία ερώτηση μόνο για να δείξω το ενδιαφέρον μας. Στην Κροατία, όταν είχα πάει με μια αντιπροσωπεία, Καλά, ούτε ερώτηση να κάνω <laughs> λοιπόν. Υποστηρίζω, δεν έχω χρόνο ούτε να κάνω αυτή την ερώτηση. Ε, εκφράζω την υποστήριξη ε, στη δραστηριότητά σας. Η κυρία Μπρισάζη, τελευταία ε, συνάδελφος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω την ευκαιρία να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Ε, δεν θα επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν. Θα ήθελα να ε, καλέσω την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή και να την εγγράψουν ε, σε μια ημερήσια διάταξη ως μοναδικό σημείο να αφιερώσουμε μια ολόκληρη συνεδρίαση σε αυτό. Είδατε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα, χρειάζεται και αξίζουν χωριστή συζήτηση. Εγώ είμαι πρόσφυγας από τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ε, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, εκπροσωπώ τη Σουηδία όπου και έχω εκλογεί και θα ήθελα όμως να τονίσω όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και σε ξεχωριστή ακρόαση να ασχοληθούμε μόνο θεματικά με αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σκούκαν. Ήταν τελευταία παρατήρηση, παρέμβαση. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Ε, όσοι θέλετε να συναντήσετε τους προσκεκλημένους μας, θα έχετε την ευκαιρία να τους δείτε από τις 2 μέχρι τις 3. Θα είναι στη διάθεσή σας στην αίθουσα Πόλα Ρίσπακ 6Β1, στον έκτο όροφο, HS6B. Ε, b πολύ, Πρόεδρος. Θα ήθελα να σας πω μόνο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο σας για σας, αλλά και για μας. Είναι πρότυπο για να δούμε πώς ε, τέτοιες περιφέρειες που έχουν πληγεί ε, από πολλά δεινά κάνουν τη μετάβασή τους. Σήμερα το απόγευμα θα συζητήσουμε τη μετάβαση στην Αργεντινή. Γι' αυτό θα ήθελα να διδαχτούμε από ε, τη δική σας ενότητα πώς καταφέρατε να την οικοδομήσετε, ενωθείτε μεταξύ σας μετά από τόσο πικρές και δυνηρές εμπειρίες και θα αποτελέσει αυτό και δίδαγμα για άλλους. Ευχαριστώ. Διακόπτε τη συνεδρίαση συνέχεια στις 3, διευρυμένο προεδρείο στις 2 εδώ. Καλή επιτυχία.